Έχουμε ένα σημαντικό θέμα σήμερα. Γεωργία και κλιματολογικές αλλαγές. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν εδώ και πολύ καιρό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να μελετήσουμε σε βάθος αυτό που όλοι πιστεύουμε ότι η γεωργία είναι τμήμα του προβλήματος αλλά σίγουρα είναι και τμήμα της λύσης του προβλήματος. Καλωσορίζω τους εμπειρογνώμονες που έχουμε καλέσει. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς Ήρθατε από πολύ μακριά για να μεταφέρετε τις γνώσεις σας στη συζήτησή μας για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και τις κλιματολογικές αλλαγές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας. Πάρα πολύ σύντομα θα γίνει μία από τις βασικές προκλήσεις της ΚΑΠ, η κλιματολογική αλλαγή. Και θα πρέπει από τώρα να προσπαθήσουμε να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στη Γεωργία, να προσαρμόσουμε τις ανάγκες των γεωργών στις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν ε, ξεκινήσει και να μειώσουμε γενικότερα τις εκπομπές. Πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση, έχει αργήσει. Παράλληλα, με τις σκέψεις τις οποίες κάνουμε για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2013. Το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών δεν έχει εξεταστεί σε βάθος. Η κλίδα των αλλαγών που είναι απαραίτητες για τη γεωργία βρίσκονται στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε φόρος ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, βλέποντας ακριβώς τα προβλήματα που δημιουργούν οι κλιματολογικές αλλαγές, και ποιες είναι οι προσδοκίες των πολιτών από το κομμάτι της γεωργίας θα πρέπει να στρέψουμε τις απαιτούμενες και δίκαιες θα έλεγα μορφές χρηματοδότησης στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ εκεί που χρειάζεται. Και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Στεφάν Λεφόλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και εσείς και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ και ιδίως ε, όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ να συμμετάσχουν στις συζητήσεις μας. Όπως ε, το είπε ήδη ο πρόεδρός μας, πιστεύω ότι η υπερθέρμανση του κλίματος είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο σήμερα από πολιτική άποψη, ιδίως μετά την αποτυχία της Κοπενχάγης. Και λέω αποτυχία της Κοπενχάγης και ταυτόχρονα πιστεύω ότι η Κοπενχάγη ε, θα μπορούσε να είναι μια ήταν μια σημαντική στιγμή γιατί όλες οι μεγάλες χώρες του κόσμου ε, βρέθηκαν γύρω από ένα τραπέζι για να συζητήσουν το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Θεωρώντα δηλαδή ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα. Ναι, μεν οι λύσει δεν βρέθηκαν, αλλά η συνειδητοποίηση των ε, προηγμένων χωρών και των αναδιόμενων χωρών που γνωρίζουν σήμερα μια ταχεία οικονομική εξέλιξη το σύνολο του κόσμου συνειδητοποίησε λοιπόν την ανάγκη να επεξεργαστούν κάποιες λύσεις για να καταπολεμήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό η γεωργία όπως υπόθηκε προηγουμένως είναι, ήταν ταυτοχρόνως ένας παράγων της ε, θέρμανσης, υπερθέρμανσης του κλίματος και θα πρέπει μελλοντικά να είναι ένας παράγων ο οποίος θα είναι σε θέση να επιφέρει κάποιες λύσεις στον αγώνα αυτό κατά της υπερθέρμανσης του κλίματος. Αυτό είναι ένα πρώτο μήνυμα λοιπόν, το μήνυμα ότι η γεωργία ε, φύση, δηλαδή μέσω της σχέσης με το έδαφος, με τους ζώντες οργανισμούς, είναι ένας μείζον παράγων ο οποίος θα πρέπει να κινητοποιηθεί ούτω ώστε να υπάρξει μια αλλαγή στο μοντέλο της εξέλιξης έτσι όπως το γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Της ανάπτυξης μάλλον έτσι όπως το γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Το λέω γιατί η υπερθέμανση του κλίματος δεν ε, μπορεί να περιοριστεί στους δύο ε, βαθμούς Κελσίου. Ε, όπως συνήθω προσδιορίζεται. Θα έλεγα ότι στι ε, απαρχέ του 21ου αιώνα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι φυσικοί πόροι, οι πόροι σε ορυκτά καύσιμα έχουν όλοι όρια. Και αν μέχρι τώρα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι, θα, ότι μπορούμε να αναπτυσσόμεθα καταναλώνοντας όλους αυτούς τους πόρους, όλα αυτά τα αποθέματα, σήμερα πλέον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να συνειδητοποιήσουμε ότι χρήζουν μιας διαχείρισης και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον αν θέλουμε να εγγυηθούμε ένα μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το διακύβευμα Δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε την ιδέα ότι δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη εις βάρος της φυσικής ισορροπίας και της ισορροπίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του πλανήτη. Και αυτό σχετίζεται με το θέμα της υπερθέρμανσης του κλίματος, αλλά σχετίζεται με όλα τα άλλα θέματα, όπως είναι το θέμα των υδάτων, που θα έχει μείζωνα σημασία στο μέλλον, και σκέφτομαι επίσης το θέμα του εδάφους, γιατί γνωρίζουμε ότι σήμερα ε, πάση επίση υφίσταται αρνητικέ επιπτώσει από ένα μοντέλο ανάπτυξη. Έχουμε τα φαινόμενα ξηρασία, για παράδειγμα. Πρόκειται λοιπόν για μια ανάπτυξη στην οποία θα πρέπει, την οποία θα πρέπει να επηρεάσουμε μέσω τη γεωργία και τη χάραξη μια νέα πολιτική, η οποία να λαμβάνει υπόψη το σύνολο του θέματο, όλε τι πτυχέ του ζητήματο. Και τώρα φτάνω στι απαντήσει και στην έκθεσή μου. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι θα ήθελα να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε την πολιτισμική αλλαγή που είναι αναγκαία ούτε ώστε να προσεγγίσουμε σωστά αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα και η Επιτροπή Γεωργίας καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίσουν τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη γεωργία κάνοντας μια διάκριση μεταξύ των προβλημάτων, ξεχωρίζοντας τα προβλήματα. Δηλαδή, για το κάθε πρόβλημα υπάρχει μια οδηγία. Οδηγία για τα εντομοκτώνα, οδηγία για το έδαφος, οδηγία για τα ύδατα ε, οδηγία για την ευημερία των ζώων, κάτι που συζητήσαμε χθε. Και κάθε φορά υπάρχει μια οδηγία, ένα σύνολο κανόνων και διατάξεων που θέλουμε να τηρούνται και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τους ε, αγρότες και ε, συσσωρεύονται. Ε, και τελικά στο τέλος οι στόχοι που θέτουμε γίνονται, δεν είναι πλέον εύληπτοι και δυσχεραίνουν το βίο των αγροτών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά, τους ώστε να ευθύσουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Αυτό αποκαλείται συστημικό μοντέλο προσέγγισης. Η γεωργία εντός ενός οικοσυστήματος είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να προσληφθεί στη σφαιρικότητά του και θα πρέπει να πάψουμε να ξεχωρίζουμε τους τομείς για να θεσπίσουμε κάποιες οδηγίες που καλούμεθα να εφαρμόσουμε στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε για πρώτη φορά να ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία προσεγγίζει με σφαρικό τρόπο το θέμα. Η κλιματική υπερθέρμανση μας υποχρεώνει να προβληματιστούμε σε σχέση με δύο στοιχεία. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την κατανάλωση και τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση κλειδί. Και δεύτερον, πώς η γεωργία μπορεί η ίδια να συμμετάσχει στην ε, αποθήκευση στοιχείων των αερίων ε, ε, θερμοκηπίου, ιδιαίτερα του άνθρακα μέσω ενός νέου μοντέλου σκέψης. Δηλαδή, από τη μία να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων, από την άλλη να προσπαθήσουμε να δεσμεύσουμε ένα μέγιστο, μια μέγιστη ποσότητα του άνθρακα στο έδαφος. Το έδαφος περιέχει 70 δισεκατομμύρια τόνους ε, άνθρακα ε, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό και μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την απόδοση. Γιατί λέω ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα συστημικού χαρακτήρα, γιατί εάν υιοθήσουμε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση θα πρέπει να υιοθήσουμε κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι να μας επιτρέπουν να καταλώνουμε λιγότερη ενέργεια, να εκπέμπουμε λιγότερα αερία θερμοκηπίου έχοντας σαν στόχο ταυτόχρονα τη διαφύλαξη του εδάφους, των υδάτινων πόρων επίσης και να επιτρέπουμε στο έδαφος να δεσμεύει ένα μέρος του άνθρακα και εν πάση περιπτώσει να το διαφυλάσει, να το διατηρεί. Το δεύτερο στοιχείο είναι να προσπαθήσουμε να προβληματιστούμε για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα και με έναν ε, βέλτιστο τρόπο ε, τη φύση σε αυτά που μας προσφέρει και σκέφτομαι με αυτό, εννοώ με αυτό την ηλιακή ενέργεια τη φωτοσύνθεση. Η γεωργία διαχειρίζεται ακριβώς τη φωτοσύνθεση, ένα φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, που μας επιτρέπει να μετατρέψουμε τη λαϊκή ενέργεια σε βιομάζα, σε ενέργεια, σε άνθρακα, να δημιουργήσουμε ζωή να ζωγονίσουμε το έδαφο. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό θέμα. Και αυτό λοιπόν το οποίο προτείνω στην έκθεσή μου είναι να πάρουμε όλα τα στοιχεία που μα επιτρέπουν να συνδυάσουμε ταυτόχρονα ε, τη μείωση της κατανάλωσης ε, ορυκτών πηγών, μείωση εκπομπών αερίων θερμοκήπιου, έχοντα σαν στόχο να εξασφαλίσουμε μια δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα μέσω των γεωργικών καλλιεργιών. Αυτός είναι, αυτό είναι το αντικείμενο της έκθεσής μου. Και ε, σκέφτομαι ότι στις προηγούμενες εκθέσεις ε, και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά στοιχεία στο τραπέζι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα συγκεντρώσουμε, να τους προσδώσουμε ένα νέο νόημα και μια συνοχή. Και εγώ θέλω να προσπαθήσω να προτείνω ακριβώς μια σφαιρική προσέγγιση της εξέλιξης της γεωργίας που ξεκινάει από την βιολογική γεωργία, η οποία υπάρχει και μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός στόχος ε, που προσδιορίζουμε. Θα πρέπει να έχουμε έναν πλατύτερο στόχο που αφορά το σύνολο της γεωργίας, ώστε να εξασφαλίσουμε μια μετάβαση στη γεωργία από το συμβατικό μοντέλο προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής που λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον ε, και μάλιστα με έναν οικονομικά βιώσιμο τρόπο γιατί είμαστε σε ένα κόσμο που δεν ε, είμαστε μόνοι μας και θα πρέπει να έχουμε και αυτή την οικονομική διάσταση κατά νου γιατί πραγματικά καθορίζει το σύνολο των γεωργικών δραστηριοτήτων. Στην έκθεσή μου έκανα ορισμένε προτάσει, συμπεριέλαβα κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν στι συζητήσει και προσπάθησα να τα συγκεντρώσω για να ε, ανοίξω προοπτικέ σε μια νέα γεωργική πολιτική γιατί στην ουσία εάν ευθύσουμε αυτό το διάβημα θα πρέπει στη συνέχεια να μπορεί να μεταφράζεται σε μια γεωργική πολιτική η οποία να επιτρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή τη σφαιρική μετάβαση, να αναγνωρίσουμε για τον γεωργό όχι μόνο τον κοινωνικό του ρόλο, ε, διατήρησης της ε, ε, ποικιλομορφίας στη διαχείριση των καλλιεργικών αλλά επίσης την ε, σχέση με τη διαφύλαξη του και η προστασία του εδάφους. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και πραγματικά συγκέντρωσα πολλά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη βιολογική γεωργία αλλά και στις νέες τεχνικές, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε εδώ και ήρθαν εδώ πολλοί εμπειρογνώμονε για να μα δείξουν ακριβώ τι συμβαίνει, Νέε τεχνικέ που επιτρέπουν να συνδυάσουμε τα τρία ή τέσσερα στοιχεία τα οποία προανέφερα, ε, δέσμευση του άνθρακα, μείωση τη κατανάλωση τη ορεικτή ενέργεια προστασία των φυσικών πόρων. Και εν κατακλείδη λοιπόν, γιατί ήδη μακρηγόρησα, αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι σε σχέση με το ερώτημα που τίθεται για την κλιματική υπερθέρμανση θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιους προβληματισμούς εν σχέση με τη διατύπωση μιας γεωργίας η οποία από οικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη να είναι αποδοτική και στους τρεις αυτούς τομείς και η Ευρώπη να διαδραματίσει ένα μείζωνα ρόλο σε ολόκληρο τον κόσμο σε σχέση με το θέμα αυτό. Το γνωρίζουμε λοιπόν, τα διατροφικά, το διατροφικό ζήτημα είναι ένα ουσιαστικό θέμα, ένα δισεκατομμύριο ανθρώπινα όντα υποφέρουν από πείνα ε, ε, στη διάσκεψη της ε, Κοπεχάγης υπάρχει από τη μία πλευρά έχουμε φαινόμενα ξηρασίας, από την άλλη έχουμε φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες και θα πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι, επειδή ακριβώς οι αγρότες μας έχουν μια ιστορία, ένα πολιτισμό πίσω τους και είναι σε θέση να εφαρμόσουν κάποιες ισορρευμένες εμπειρίες. Θα πρέπει εμείς λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτή τη μετάβαση η οποία θα καταστήσει την Ευρώπη ένα παράδειγμα σε πλανητική κλίμακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Στεφάν, τον ευχαριστώ για τις απόψεις που εξέφρασε και για τη σφαιρική αντίληψη που μας προτείνει να έχουμε γύρω από το θέμα. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τη σειρά των εμπειρογνωμόνων με τον κύριο Ντόναλ Ρισκόνσκι από το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το USDA. θα μας μιλήσει για τις πρακτικές λύσεις και τις δυνατές πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του περιορισμού του διοξιδίου του άνθρακα στο έδαφος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεφόλ ε, έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή Οπότε υπάρχει μια κατανόηση για την ανάγκη αυτών των πληροφοριών σε σχέση με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Παγκόσμιες οι ανησυχίες. Χρειάζεται λοιπόν κάποια μορφή αηφόρος γεωργία. Πρέπει να μας απασχολήσει η οικονομία, η ασφάλεια των τροφίμων, πτυχές της κλιματικής αλλαγής, βιοενέργεια, ανανεώσιμη ενέργεια και εμείς εξαρτώμεθα και από το πετρέλαιο, από το εξωτερικό. Επίσης η περιβαλλοντική ποιότητα είναι σημαντική. Όλα αυτά ανάγονται στη διαχείριση εμέ του άνθρακα. Συγκεκριμένο παράδειγμα ε, είναι η διατήρηση του εδάφους σε σχέση με την αηφόρο γεωργία. Και εδώ όλα εξαρτώνται από τον άνθρακα και μίσε. Θέλουμε την καλύτερη διαχείριση άνθρακα στο έδαφος που μπορούμε. Η αηφόρο γεωργία απαιτεί διαχείριση του κύκλου του άνθρακα και οι υπηρεσίε οικοσυστημάτων ε, είναι υπεύθυνε για τη διαχείριση του κύκλου του άνθρακα. Όπως ανέφερε ο κ. Λεφόλ, η παγίδευση γίνεται ω επιτοπλίστων στα πλαίσια τη φωτοσύνθεσης και αυτή την ενέργεια τη χρησιμοποιούμε για την ε, ε, σε τρόφιμα. Η αντίστροφη ε, ε, διαδικασία της φωτοσύνθεσης είναι η εξατμισιοδιαπνοή που μας επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας και συνέχεια φυσιολογικών λειτουργιών. Εκλείεται ενέργεια έτσι Όλες αυτές οι λειτουργίες όμως ε, ε, έχουν σχέση με τη διαχείριση του άνθρακα. Πολλοί υποσυτίζονται, ε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κλιματικά στον πλανήτη, μας ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών μας και υπάρχει μια δυνατότητα διατήρησης του συστήματος που είναι η γεωργία συντήρησης, διατήρησης που εξαρτάται από το έδαφος όπου ζούμε το ζωντανό ε, έδαφος που εξαρτάται πάλι από τον άνθρακα. Οπότε η συνιστόσα κλειδί εδώ είναι η διαχείριση του άνθρακα κοντά στην επιφάνεια των εδαφών μας. Όλοι θέλουμε υψηλή ποιότητα ζωής και εξαρτώμεθα από τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων τα, οι περισσότερες υπηρεσίες οδηγούν σε αυτήν την γεωργία διατήρησης που απαιτεί λιγότερο ε, ε εντατική ε, άρρωση. Ε, ο οργανικός άνθρακας είναι σημαντικός στο έδαφος και πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό το υλικό. Στα συστήματα διατήρησης γεωργίας ε, χρησιμοποιούμε την ελάχιστη άρρωση, ελάχιστη διατήρηση χάραξη του εδάφους. Ε, επίσης έχουμε άμυψη σπορά, επισπορά, άλλου είδους διακαλλιέργειες. Επίσης ε, χρησιμοποιούμε τις έννοιες ε, της συνεχιζόμενης κάλυψης απορριμμάτων ή πολυμάτων. έτσι λοιπόν θα ήθελα να γίνει κατανοητό ότι ο άνθρακας είναι το C από το carbon που από το C αρχίζει και η λέξη conservation διατήρηση. η βιομάζα ε, έχει σχέση με τον άνθρακα. Η διάβρωση επίσης, ε, αν δούμε συστήματα χωρίς άρρωση ε, με απορρίμματα στην επιφάνεια, πάλι επηρεάζονται από τον άνθρακα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι η πραγματική διατήρηση είναι η διαχείριση του άνθρακα και η διατήρηση μπορεί να είναι από τα πρώτα βήματα για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικός ο άνθρακας για μας, είναι το κέντρο αυτού του μαγικού τριγώνου του εδάφους. Υπάρχει βιολογική, υπάρχουν βιολογικές, φυσικές, χημικές διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές και μικρή ποσότητα άνθρακα είναι σημαντική για να διατηρηθούν οι κρίσιμες λειτουργίες του εδάφους που προϋποθέτουν την παραγωγή καλλιεργιών και την ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι λοιπόν ο κύκλος του άνθρακα είναι η βάση της ζωής μας, της επιβίωσής μας, της ε, παραγωγής ε, τροφίμων για τον κόσμο, διατήρηση ε, επίσης της λειτουργίας του εδάφου και των μικροοργανισμών εκεί. Ο αέρας, το νερό είναι σημαντικά για τη φωτοσύνθεση και την συλλογή ενέργειας για τη δική μας χρήση όπως επίσης και για τη μικροβιολογία του εδάφους που είναι τόσο πολύ σημαντική για μας. Οι δυο διαδικασίες που εμείς στη Γεωργία θα πρέπει να διαχειριστούμε είναι η φωτοσύνθεση και η διαπνοή. Σημαντικό είναι να είναι αυτές οι διαδικασίες όσο γίνεται πιο αποτελεσματικές και να αντιμετωπίζουν επίσης και τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το φυτό άνθρακα γιατί ε, αν το δούμε έτσι θα δούμε διαφορετικά και τη, το, τη διατήρηση, συντήρηση. 45% πολλών φυτών αποτελούνται από άνθρακα. Έτσι λοιπόν έχουν ε, κάποια ισχύ. Το παγιδεύουμε, τον άνθρακα, τον αποθηκεύουμε, υλικό βιομάζας και ε, έχουμε πηγή τροφίμων επίσης εκτός από αποθήκευση ενέργειας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εισρωή άνθρακα του εδάφους. Η έχουμε περιβαλλοντικά ωφέλη από τη διαχείριση του άνθρακα, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για μας. Όλα αυτά συμβάλλουν σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής για μας. Αν σκεφτόμαστε λοιπόν τα φυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε ε, ως ε, άνθρακα και όχι κατάλοιπα φυτών ε, ή απορρίμματα φυτών. Όταν αξιοποιήσουμε αυτές, αυτούς τους πόρους στην γεωργία τα, ε, οι υπηρεσίε οικοσυστημάτων ε, περιστρέφονται γύρω από τον άνθρακα. Τα τρόφιμα, οι ζωοτροφέ, οι ίνες ε, και τα βιοκαύσιμα τώρα όλα ρυθμίζονται από αυτό τον κύκλο του άνθρακα. Και όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε να διαχειριζόμαστε σωστά τον κύκλο, τόσο καλύτερα θα είναι για τις μελλοντικέ γενναίες. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία συντήρηση διατήρηση και την παγίδευση δέσμευση του άνθρακα, πολλά συζητούνται τώρα σε σχέση με τα ωφέλη που μπορεί να αποδοθούν σε αυτό. Ω παράδειγμα χρησιμοποιώ κάποια δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στι ΗΠΑ και δείχνουν ότι υπάρχει κάποια παγίδευση δέσμευση άνθρακα στα επιφανειακά στρώματα του εδάφου. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση. στι ΗΠΑ έχουμε 16.000 διαφορετικά εδάφη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, κάνουμε συγκρίσει στα οικοσυστήματα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι δύο βασικές παράμετροι σε ένα βιολογικό σύστημα είναι η θερμοκρασία και η βροχόπτωση που παρατηρούνται στα διαφορετικά οικοσυστήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και για τις μέσες τιμές υπάρχουν τεράστιες διακυμάνσεις. Σε επιστημονικό επίπεδο λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις ε, ε, βάσιμες. Όμως υπάρχει γενικότερη συσσόρευση ε, άνθρακα στα συστήματα διατήρησης που πρέπει να γίνουν κατανοητά από τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Στις ΕΠΑ υπάρχουν περισσότερες από 150 εθελοντικές αγορές άνθρακα. Υπογραμμίζω τη λέξη εθελοντικές γιατί συμβάλλουν στην κατανόηση της εμπορίας του άνθρακα όμως ε, δεν ε, υπάρχει πρόσθετη αξία εδώ γιατί δεν υπάρχει ακόμα στη ΣΥΠΑ πολιτική αλλαγής του κλίματος. Ε, όμως θα επηρεαστεί το μέλλον του προγράμματος για την αλλαγή του κλίματος και η έκβαση βεβαίως της ε, Συνόδου Κορυφής της Κοπενχάγης άφησαν κάποια βεβαιότητα. Όμως νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην μείωση της φτώχειας. Θα έχουμε περισσότερη ε, βιώσιμη ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη, ασφάλεια τροφίμων και ενέργειας και βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν ε, ισχύει ένα μέτρο για όλα τα προβλήματα, ε, διότι υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα στα συστήματα γεωργίας. Υπάρχει μια αγορά, ε, το Chicago Climate Exchange, μια αγορά και υπάρχουν πάρα πολλά ε, offsets, αντισταθμίσεις που μπορείτε να δείτε. Ε, το ένα είναι του άνθρακα του εδάφους και βλέπουμε το, τους μετρικούς τόνους αλλά και την αξία όλων αυτών των τύπων αντισταθμίσεων για την καλύτερη διαχείριση του άνθρακα. Υπάρχουν και άλλες αντισταθμίσει στη γεωργία, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ στο αντισταθμίση, στην αντιστάθμιση του ε, άνθρακα του εδάφους. Υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές, όχι τόσο ριζικές όσο θα θέλαμε, αλλά μπορεί να υπάρξει ε, αυξανόμενη αξία σε σχέση με αυτά τα προγράμματα. Έχω ένα παράδειγμα ε, μιας ε, προβολής σε σχέση με την αξία της αγοράς άνθρακα το 2012 και ε, η αξία έχει υπολογιστεί ως 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, είπα, είναι πάρα πολλά χρήματα και ε, αυτό είναι ε, όχι προσωπική μου ε, πρόβλεψη αλλά ε, μία πρόβλεψη πιο επίσημη. Εάν το πολλαπλασιάσετε θα, με το, θα, μπορείτε να υπολογίσετε την αξία σε ευρώ επίσης και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αυτήν την εξέλιξη. Όμως θα πρέπει κάποια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα να τα δούμε σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ως επιστήμον όμως θα πρέπει να, δώσω κάποια να σας δώσω τα θετικά στοιχεία που αφορούν την παγίδευση του ε, άνθρακα. Τα... Οι υπηρεσίε οικοσυστήματος ε, είναι ακτίνες που βγαίνουν από τον βασικό ε, πυρήνα του άνθρακα. Είναι ο, ο, ο άνθρακας ε, ο, το βασι, βασικός άξονας αυτής αυτού του τροχού ε, οι υπηρεσίε οικοσυστήματος μπορεί να συμβάλλουν λοιπόν σε ό,τι χρειάζεται για τα γεωργικά συστήματα, δηλαδή αυξημένη ικανότητα διατήρησης, συγκράτησης του ύδατος, ε, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα χρήσης Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ωφέλη για τα γεωργικά συστήματα παραγωγής ώστε να είναι αηφόρα, βιώσιμα. Υπάρχει κάποια αυξημένη βιοδραστηριότητα, ε, ε, υπάρχουν περίπου 13 τέσσερα ωφέλη που αναγράφονται εδώ που μπορεί ε, μεμονωμένα να μην ε, έχουν μεγάλη συμβολή αλλά συλλογικά επηρεάζουν, ε, όλα μαζί επηρεάζουν πολύ το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, αν δούμε ότι ο πυρήνας, ο βασικός, το, το, το αξόνιο είναι ο άνθρακας, τότε μπορούμε ανάλογα να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας. Και θα ήθελα στο τέλος να δείξω αυτή τη διαφάνεια ε, σχετικά με το αποτύπωμά μας σε άνθρακα. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται και τα παιδιά ε, για να προετοιμάζονται. Ε, θα πρέπει το αποτύπωμα του άνθρακα να είναι μικρό και θα πρέπει ο άνθρακας, τον άνθρακα να τον διαχειριζόμαστε για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρεϊντκόσκι. Ας περάσουμε λοιπόν στην επόμενη παρουσίαση. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες γενικά παρουσιάσεις σήμερα, είμαι βέβαιος. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Φρανκομάρα, διευθυντή έρευνας του Τιγασκ. Θα μας μιλήσει για τις λύσεις που υπάρχουν για τη μείωση των ε, αερίων του ε, θερμοκηπίου για τα μυρικαστικά. Ο κύριος Σομάρα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής και εσάς για την δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω το λόγο στα θέματα των κλιματολογικών αλλαγών και της γεωργίας. Θα μιλήσω για τη μείωση της εκπομπής αερίων από τα μυρικαστικά. Θα ήθελα να σας υπογραμμίσω κάποιες από τις τεχνολογίες οι οποίες είναι διαθέσιμες ή θα είναι διαθέσιμες για τη μείωση αυτή. θα δούμε από πού προέρχονται καταρχάς αυτές οι εκπομπές των μυρικαστικών. Εδώ βλέπετε την εικόνα, αν θέλετε, της εκπομπής αυτών των αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι η εντερική ζήμωση που προέρχεται από την κτηνοτροφία αφορά περίπου το 1 τρίτο γενικά των εκπομπών της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα είναι 20% και φυσικά υπάρχει και το θέμα της ποιότητας της, ε, της γης η οποία δεν ξεπερνάει το 20% επίσης. Και εκεί τίθεται το θέμα της διαχείρισης του διοξιδίου του θείου. εν μέρη προέρχονται επίσης και από την εναπόθεση ε, των ούρων των μυρικαστικών στις ε, καλλιεργούμενες επιφάνειες ή στις επιφάνειες βοσκής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι ε, των εκπομπών στο πρωτοξίδιο του άξε, πρωτοξίδιο του θείου προέρχονται από τα μυρικαστικά, σχεδόν το 50% αν δει κανεί ποιε είναι οι προοπτικέ για τι εκπομπέ αυτέ στο μέλλον, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαφορετικέ τάσει τα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Οι εκπομπές στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες είναι πλέον στάσιμες και εξακολουθούν να είναι στάσιμες τις τελευταίες δεκαετίες και η προοπτική επίσης δεν προβλέπει αλλαγές για την επόμενη δεκαετία ενώ στις αναπτυσσόμενες περιοχές αυξάνονται σημαντικά οι εκπομπές από τις γεωργικές περιοχές γιατί αυξάνεται η παραγωγή στις χώρες αυτές πάντα για να έχουμε μια σφαιρική προοπτική σχετικά και με τις δυνατότητες αντιμετώπισης και μετριασμού του φαινομένου. Εδώ βλέπετε μια διοφάνεια από ε, το, την έκθεση του IPCC του 2007 για τις σφαιρικές δυνατότητες μετριασμού των συνεπειών στην Γεωργία. Η έκθεση του IPCC λέγει ότι υπάρχουν δυνατότητες για μετριασμό, ελάφρυνση δηλαδή του φαινομένου αυτού μέσω της σωστής ε, διαχείρισης του άνθρακα που βρίσκεται, που εναποτίθεται στο έδαφος. Αν πάρετε τη δεύτερη από το τέλος στήλη θα δείτε τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από την κτηνοτροφία θα δείτε ότι από τις δυνατότητες μετριασμού εκεί το ποσοστό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Η γεωργία γενικά μπορεί να συνεισφέρει κατά πολύ. Όχι ασήμαντο το ποσοστό βέβαια το οποίο προέρχεται από την κτηνοτροφία, αλλά όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής έχουμε να κάνουμε με μικρές δυνατότητες αλλαγής της κατάστασης και εκθέσεις από διάφορους γεωργικούς οργανισμούς λέγουν ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες βελτίωσης των γεών για την ε, μείωση γενικά της εκπομπής αερίων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να μειώσουμε ακριβώς αυτή την εντερική ζήμωση. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες στη διάθεσή μας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και υπάρχουν πολλές, πολλά καλά υποσχόμενες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές, όπως η αντικατάσταση της ακατέργαστης χορτονομής, η συμπλήρωση με οργανικά οξέα, η προσθήκη λιπιδίων στην δίαιτα των ζώων, η μονενσίνη, νατριούχος μονενσίνη την οποία μπορούμε να δώσουμε στα ζώα και η οποία βελτιώνει την κατάσταση. Η βελτίωση επίσης των περιοχών όπου εκτρέφονται τα ζώα, όπως επίσης και η συμπερίληψη λαχανικών στην τροφή. Υπάρχουν γενικά αρκετά μέτρα τα οποία είναι γνωστά σε αυτή τη φάση και μπορούν να βοηθήσουν τη μείωση των εκπομπών από τα μυρικαστικά. Το θέμα είναι ότι αυτές οι μέθοδοι σε αυτή τη φάση δεν είναι ιδιαίτερα οικονομικά ελκυστικές. Η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών χωρίς κίνητρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα. Κάποιες από τις ε, ε τεχνολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα βράχυπρόθεσμες μπορεί σε πειραματικό στάδιο να είναι πολλά υποσχόμενες όπως είπα αλλά αν εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα δεν ξέρουμε ακριβώς τι αποτελέσματα θα δώσουν και απαιτείται πολύ μεγαλύτερη έρευνα πριν σταθούμε ικανοί να εφαρμόσουμε τις μεθόδους αυτές σε ευρύτατα πλαίσια. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε και θα επανέλθω στις τεχνολογίες τις οποίες είπα προηγουμένως. Υπάρχουν άλλα θέματα που κάνουμε στη Γεωργία τα οποία βοηθούν στη μείωση της εκπομπής αερίων. Το βασικό είναι η βελτίωση στην παραγωγικότητα που χαρακτηρίζει την γαλακτοτροφία την ευρωπαϊκή τα τελευταία 20-30 χρόνια αυτή η βελτίωση στην παραγωγικότητα αποτελεί μια πάρα πολύ στρατηγική για μας για τη μείωση των εκπομπών ανά κιλό προϊόντος. Και μιας και έχουμε να κάνουμε με ένα πλαίσιο αγοράς το οποίο θα επιζητεί περισσότερες τροφές από ό,τι σήμερα, περισσότερες ποσότητες τροφές, και μιας και δεν έχουμε άλλες μεθόδους, καλό θα είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στη μείωση των εκπομπών ανά κιλό προϊόντος το οποίο θα παράγουμε. Όταν βλέπει κανείς την Ευρωπαϊκή Γεωργία για την εκπομπή μεθανίου ανά κιλό γάλακτος σαν παράδειγμα, βλέπουμε ότι τα πάμε αρκετά καλά σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Και έχει βελτιωθεί η εκπομπή μεθανίου τα τελευταία 20 χρόνια, έχει μειωθεί δηλαδή. Στη δική μου χώρα, στην Ιρλανδία, σαν παράδειγμα, ανακυλό το 1990 αν το συγκρίνει κανείς με το 2006 υπάρχει μια μείωση κατά 13% ανακυλό γάλακτος. Αυτό δεν σας φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικό το ποσοστό και αν συγκρίνει κανείς το τι συμβαίνει με άλλες χώρες, αν δει κανεί το τι συμβαίνει στη Νέα Ζηλανδία ή στις Ηνωμένε Πολιτείε, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη εκεί μείωση. Γιατί οι ποσοστώσεις τις οποίες είχαμε ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τα τελευταία χρόνια είχαν τελικά σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κέρδους από τη βελτίωση της παραγωγικότητας την οποία ταυτόχρονα πετύχαμε. Επίσης το θέμα των ζωοτροφών. Εκεί πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος και πρέπει να ανοίξουμε νέους δρόμους θα έλεγα σε επίπεδο ζωοτροφών και στη διατροφή των ζώων γενικότερα. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Βέβαια οι αλλαγές είναι ριζοσπαστικές τα τελευταία 30-40 χρόνια, αλλά για τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα μείωσης Ε, όπως ακριβώς σας έδειξα και στις προηγούμενες διαφάνειες. Αυτή είναι μια τάση η οποία θα συνεχιστεί και αναφέρομαι πάντα στη μείωση του μεθανίου. Έχουμε αρχίσει επίσης ε, να ε, ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα για εκτροφή ζώων που έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και σε σχέση με την κατανάλωση τροφών, κτηνοτροφών και πρέπει αυτά να τα συμπεριλάβουμε στα προγράμματα εκτροφής. Με λίγα λόγια πρέπει να χρειάζεται λιγότερη τροφή για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας του τελικού προϊόντος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μείωση του μεθανίου με αύξηση ή διατήρηση των ιδίων επιπέδων παραγωγής γάλακτος. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ αρχικά στάδια της ε, παραγωγής αυτής. Ε, υπάρχει η δυνατότητα με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε να πούμε ότι κάποιες ποικιλίε ζώων παράγουν λιγότερο μεθάνιο από ότι κάποιες άλλες ε, ποικιλίε. Αυτό ίσως είναι ένα γενετικό χαρακτηριστικό των ζώων. Αν εντοπίσουμε σωστά τις κατηγορίες αυτών των ζώων, και αν μπορούμε να επιλέξουμε ακριβώς ε, κάποιες ποικιλίε ζώων οι οποίες παράγουν χαμηλά επίπεδα ή χαμηλότερα εν πάση περιπτώσει επίπεδα μεθανίου αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Βέβαια είναι πρώιμη η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα έχουμε όμως προοπτικές. Και τέλος σε σχέση πάντα με την εταιρική ε, ζήμωση να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο οι τεχνολογίες μέχρι τώρα δεν έχουν πετύχει πάρα πολλά σε επίπεδο μείωσης του μεθανίου είναι το ότι δεν κατανοούμε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία αυτή επιστημονικά. Δεν την ελέγχουμε και δεν μπορούμε συνεπώς να πούμε ότι και οι μέθοδοι τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι αποτελεσματικές. Απαιτείται λοιπόν να ελέγξουμε με διαφορετικό τρόπο την παραγωγή προϊόντων Ξέρουμε ότι η παραγωγή μεθανίου από τα ζώα οφείλεται σε συγκεκριμένους ε, μικροοργανισμούς και στην παραγωγή αυτών των μικροοργανισμών προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε την μικροπαραγωγή των οργανισμών αυτών. Υπάρχουν ε, παγκόσμια προγράμματα γύρω από την μικροβιολογία θα έλεγα των μυρικαστικών που έχουν σαν στόχο τη μείωση ή την κατανόηση σε μια πρώτη φάση καλύτερα της διαδικασίας ε, παραγωγής ε, μεθανίου. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στο πρωτοξίδιο του θείου. Πολλές φορές ε, λέγεται ότι και εκεί είναι υπεύθυνα τα ζώα τα οποία εκτρέφουμε. Μέσω των ούρων τα οποία εναποτίθενται ε, στις ε, περιοχές όπου εκτρέφονται. Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους θα έλεγα τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ, δηλαδή για το μεθάνιο λιγότερα μπορούμε να κάνουμε, ενώ περισσότερα μπορούμε να κάνουμε για το θείο. Είναι να ελέγξουμε ακριβώς τα λοιπάσματα τα οποία χρησιμοποιούμε ε, στην παραγωγή των ζωοτροφών τις οποίες ε, ε, δίδουμε στα ζώα. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μείωση εν πάση περιπτώσει του θείου το οποίο παρέχουμε για να έχουμε και μείωση του θείου το οποίο παράγουν τα ζώα. Υπάρχουν πάρα πολλές στρατηγικές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι χρήσιμες αλλά όχι απόλυτα αποτελεσματικές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και αναστολής του θείου, μειώνουν ε, την παραγωγή θείου της περιοχές βοσκής, στα βοσκοτόπια, σε αρκετά μεγάλα ποσοστά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες όμως και σύν της άλλης το κόστος τους είναι ιδιαίτερα υψηλό 100 ευρώ ανά εκτάριο περίπου και αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε απαγορευτικό. Γίνεται μια προσπάθεια στη Νέα Ζηλανδία και το κόστος αυτό ε, υποτίθεται ότι εν πολλής καλύπτεται από την υψηλότερη παραγωγικότητα παραγωγής χορτονομής στα χωράφια στα οποία εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι αναστολής της ανάπτυξης ε, του διοξιδίου. Εν πάση περιπτώσει στην Ευρώπη σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά γιατί όπως είπα το κόστος τους είναι απαγορευτικό. Σχετικά τώρα με την, ε, ε, με την εισαγωγή λιπασμάτων και αναφέρομαι στην Ιρλανδία στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπετε ότι έχει υπάρξει μια συνεχή στάση μείωσης αμμονιούχων λιπασμάτων τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό συνδέεται με το ότι οι γεωργοί γενικά χρησιμοποιούν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο τις ζωοτροφές τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους. σχετικά με το θείο και με το πρωτοξίδιο του θείου. Οι προσπάθειες αυτές στα ε, μυρικαστικά γενικότερα δεν είναι αποτελεσματικές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το REDNEX, λιγότερο άζωτο φυσικά στα άλλη πάσματα, λιγότερο άζωτο θα υπάρχει και στην τελική παραγωγή και οι τεχνολογίες οι οποίες ε, θα χρησιμοποιηθούν και θα προέλθουν από την έρευνα η οποία γίνεται είναι νομίζω πολλά υποσχόμενες. Να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο τελευταίος ομιλητής σχετικά με τη δυνατότητα συγκράτησης του άνθρακα στο έδαφος. Υπάρχει κάποια δυνατότητα στις ε, περιοχές βοσκής των ζώων, υπάρχουν αρκετά δεδομένα τα οποία μας δείχνουν ότι συγκρατούμε στο έδαφος σημαντικά επίπεδα άνθρακα και το θέμα είναι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα έτσι ώστε να αυξήσουμε το ποσοστό συγκράτησης του άνθρακα. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την άρρωση έστω και την επιφανειακή όπου αυτό είναι δυνατό και η σωστή διαχείριση νομίζω των βοσκοτόπων μπορεί να οδηγήσει στην υψηλή συγκράτηση άνθρακα. Για να κλείσω τώρα, με τις τεχνολογίες τις οποίες έχουμε σήμερα είναι τελικά δύσκολο να μειώσουμε κάποιες ε, τις εκπομπές αυτές του μεθανίου ανακυλό του παραγόμενου προϊόντος και αναημέρα. Αλλά παρόλα αυτά η ανάπτυξη της παραγωγικότητας είναι κομβικός παράγων για την μείωση αυτή. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες σε σχέση με το πρωτοξίδιο του θείου και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε και τους τρόπους για τη συγκράτηση του άνθρακα στο έδαφος. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Υπενθυμίζω ότι μετά την επόμενη συνάντηση του κυρίου Κούκ την επόμενη παρουσίαση συγγνώμη, θα υπάρξει κάποιο σύντομο χρόνος για συζήτηση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω αν θέλετε να πάρετε το λόγο να το δηλώσετε. Μετά από άλλες δύο πάλι ε, παρεμβάσεις θα υπάρξει μια επιπλέον δυνατότητα συζήτησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να αφήσουμε στον default την δυνατότητα να ε, κλείσει τη συζήτηση. Δίνω το λόγο λοιπόν στον Ρομπ Κούκ. the land management measure policy and recommendation for the CAP. Θα κάνει συστάσεις για τις δυνατότητες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα εκ μέρους της ε, Ομάδας Πολιτικής για τη Χρήση Γης της Μεγάλης Βρετανίας να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας για να μιλήσω για το ζήτημα της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου. Η οργάνωσή μου ε, μαζί με τους ε, καλλιεργητές αναπτύσσει διάφορα αγρο περιβαλλοντικά μοντέλα στην Αγγλία. Η γεωργία συμβάλλει στο 7% του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Δηλαδή 36% των εκπομπών μεθανίου και 67% των εκπομπών πρωτοξιδίου του αζότου στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, ο τομέας διαχείρισης της γης είναι μοναδικός όχι μόνο στο ότι μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αιτίων των κλιματικών μεταβολών, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά συμβάλλοντας την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να αναπτύσσουμε κάποιου κάποιους τρόπους να εξασφαλίσουμε την διατροφική ασφάλεια, να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσουμε την αποθήκευση του άνθρακα. Και θα πρέπει να το κάνουμε διαφυλάσσοντας την φύση, η οποία είναι καθοριστική για την βιώσιμη γεωργία. Η άμβληση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί συντονισμένη δράση πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η άμβληση της κλιματικής αλλαγής είναι ένα δημόσιο αγαθό, μια υπηρεσία η οποία δεν, την οποία δεν μπορούν να παράσχουν οι ελεύθερες αγορές από μόνες τους ο πυλώνας 2 της ΚΑΠ που χρηματοδοτεί την δημιουργία δημοσίων αγαθών είναι ενδεδειγμένος για να βοηθήσει τη γεωργία να συμβάλλει στην άμβληση της κλιματικής αλλαγής γιατί παρέχει ένα ενδεδειγμένο πλαίσιο ενώ στηρίζει τις χώρες ε, μέλη για να εφαρμόσουν τοπικά τις δράσεις τους. Ο με τον πυλώνα 2 μπορούμε να εφαρρύνουμε τους καλλιεργητές να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, αλλάζοντας τη στάση τους και εφαρμόζοντας ε, νέες ε, τεχνικές. Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στην μπροστοφυλακή νέων αγροπεριβαλλοντικών μοντέλων. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να συμβάλλουμε. Πρώτον, αυξάνοντας την αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος και στις, ε, στα φυτά και μειώνοντας τις απώλειες του άνθρακα, αναβαθμίζοντας τα υποβαθμισμένα εδάφη και διαφυλάσσοντας τους τυρφώνες. Και δεύτερον, μειώνοντας το input και ε, κατευθύνοντας σωστά τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου. Ε, πολλές ε, λύσεις ε, συμβάλλουν στην άμβληση των κλιματικών μεταβολών ε, επιτρέποντας την ε, βελτίωση της παγίδευσης του άνθρακα στο έδαφος. Ε, για παράδειγμα, η δημιουργία μεμονωμένων λωρίδων εδάφους που δεν καλλιεργούνται και λειτουργούν σαν μονοτικές ζώνες. Η διαχείριση των φρακτών και η διαφύλαξη διαφόρων αρχαιολογικών στοιχείων. Εκτιμούμε ότι η μια συνδυασμένη πρόσληψη αυτών των μοντέλων αυξάνει το ποσό του άνθρακα που αποθηκεύεται στα εδάφη της Αγγλίας κατά 700.000 ε, τόνους διοξιδίου του άνθρακα το έτος. Ε, και ε, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξοικονομήσουμε σχεδόν ένα εκατομμύριο τόνους διοξίδιο του άνθρακα το έτος. Τα τελευταία τρία έτη η οργάνωσή μας δαπάνησε 90 εκατομμύρια λίρες για αγροπεριβαλλοντικά μοντέλα που οδηγούν στην άμβληση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο η εξοικονόμηση του άνθρακα ε, δεν έχει ε, σταθερό χαρακτήρα και θα μπορούσε να αναστραφεί η εξέλιξη αυτή εάν οι καλλιεργητές στραφούν σε παραδοσιακές μορφές ε, καλλιέργειας. Για παράδειγμα, εάν αρχίσουν να καλλιεργούν μια τέτοια λωρίδα γης που λειτουργεί σαν μονοτική ζώνη, τότε το, ο άνθρακας ο οποίος έχει αποθηκευτεί στο έδαφος θα απολεστεί πολύ γρήγορα στην ατμόσφαιρα. Ε, Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα από όλη τη Μεγάλη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη εν σχέση με τη χρήση της ΚΑΠ, ούτω ώστε να συμβάλλει στις ε, στην κλιματική, συνάβληση της κλιματικής αλλαγής. Στην Ουαλία έχουμε ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα ξεκινήσει το 2012 και θα εφαρμόσει μέτρα σχετικά με την κλιματική μεταβολή. Ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο βρίσκεται υπό εξέλιξη, το οποίο θα δώσει επιχορηγήσεις, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν πολλά θέματα, όπως είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ανακύκλωση των υδάτων και η χρήση πριονιδίων του ξύλου για στρομνές ζώων. Ε, τα, οι επιχορηγήσεις αυτές για την δασοκάλυψη ε, επίσης θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, Έχουμε συνείδηση ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι η μόνη χώρα που χρησιμοποιεί τα μέτρα του πυλώνα 2 για άμβληση των κλιματικών μεταβολών. Στην Αυστρία η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την αξιολόγηση του δυναμικού αποθήκευσης του άνθρακα και την ενίσχυση της περιεκτικότητας, την αύξηση της περιεκτικότητας του άνθρακα στο έδαφος μέσω διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης. Στη Γερμανία αγροπεριβαλλοντικά σχήματα, η μοντέλα συμβάλλουν στην άμβληση των κλιματικών αλλαγών, ενθαρρύνοντας τη διαφύ και την σώρευση του άνθρακα στο έδαφος μέσω νέων τεχνικών διαφύλαξη του εδάφους όπως είναι η άμεση σπορά και η δασοκάλυψη. Επίσης υπάρχει υποστήριξη για τη χρήση εξοπλισμού που βοηθάει στην διασπορά υγρής κοπριάς στα εδάφη ούτω ώστε να μειωθούν οι εκπομπέ του πρωτοξιδίου του αζότου. Στην Ιταλία ο πυλώνα 2 χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η παγίδευση του άνθρακα στα εδάφη και να δημιουργηθούν νέα δάση οι ουσιαστικές εξοικονομήσεις του άνθρακα που έχουν επιτευχθεί στην Αγγλία μέχρι τώρα είναι ένα υποπροϊόν μιας σωστής διαχείρισης που έχει άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. Η Natural England αυτή τη στιγμή αξιολογεί το πώς αγροπεριβαλλοντικά μοντέλα θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο στην κατεύθυνση της άμβλησης των κλιματικών μεταβολών προστατεύοντας και αυξάνοντας την αποθήκευση του άνθρακα. Με μια πρόθεση κάποιων εναλλακτικών λύσεων που οδηγούν στην παγίδευση του άνθρακα θα μπορούσαμε να αυξάνουμε αυτές στις δυνατότητες σημαντικά. Στην Αγγλία η υπηρεσία Environmental Stewardship ε, δεν ε, συμβάλλει τόσο πολύ στην κάλυψη γιατί εμπίπτει σε ένα διαφορετικό μοντέλο ε, ε, διαχείρισης. Άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, πολύ μεγαλύτερα αποθέματα δασοκάλυψης και έχουν καλύτερες πολιτικές διαχείρισης των δασικών εκτάσεων. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, ούτως ώστε να αυξηθεί η δασοκάλυψη και να βελτιωθεί η κατάλληλη διαχείριση των δασικών εδαφών. Ε, στην Αγγλία η κυβέρνηση πρόσφατα είπε ότι θέλει να αυξήσει την δασοκάλυψη κατά 10.000 εκτάρια το έτος για τα επόμενα 15 έτη, ούτως ώστε να παγιδευτούν 50 εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο, ε, να μπορούν να παγιδεύονται 50 εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα ανά έτος το 2050. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξουν και τα αναγκαία κονδύλια. Υπάρχει επίση μια δυνατότητα παράγοντα ενέργεια από τα υπάρχοντα δάση. Για παράδειγμα, μέχρι στιγμή 50% των δασών τη Αγγλίας δεν γίνονται αντικείμενο διαχείριση. Εάν υπάρχει στοχευμένη χρηματοδότηση, ίσω ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενεργειακών καλλιεργιών και ένα αγροπεριβαλλοντικό μοντέλο, πολλά από αυτά τα δάση θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο σωστή διαχείριση για να παραγάγουν καύσιμα από τα δέντρα, από τα δάση και μειώνοντας το, τη χρήση του άνθρακα για ενέργεια, ούτως ώστε συμβάλλοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως υπόθηκε ήδη, ε, πολλές δυνατότητες προκύπτουν από την παγίδευση του άνθρακα στο έδαφος. Ε, φαινόμενο που έχει σημαντικές συνέργειες με τη βιώσιμη ε, γεωργία και μειώνει την ευαλωτότητα σε σχέση με τις κλιματικές μεταβολές. Ε, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες όπως είναι η καλύτερη προσαρμογή στην, σε πιο υγρούς ε, χειμώνες που έχουν προβλεφθεί μελλοντικά, το οποίο σημαίνει ότι οι καλλιεργητές θα πρέπει να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ε, κοπριάς. θα μπορούσαν να σκεφτούν επίσης τη δυνατότητα αερόβιων χωνευτήρων. Επίσης η αυξημένη δασοκάλυψη θα συμβάλλει στην άμβληση των κλιματικών αλλαγών, αλλά μπορούν να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες προσαρμίσεως, για παράδειγμα ανεμοφράχτες, ούτως ώστε να υπάρχει σκιά για τα ζώα, να μειωθούν οι πλημμύρες, να μειωθεί η διάβρωση του εδάφους, να υπάρξουν ε, προστατευμένοι κότοποι για τα ζώα κλπ. Και για την παραγωγή βιομάζας βεβαίως. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα διάβρωσης, ε, ε, μείωσης διάβρωσης του εδάφους. Όλα όσα περιέγραψα περιλαμβάνει τα πολλά από τα συμπεράσματα της εξαίρετης έκθεσης του συγητού μας. Ελπίζω ότι σας έδειξα ότι στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη η δασοκομεία και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ συμβάλλουν σημαντικά στην άμβληση των κλιματικών αλλαγών. Υπό την έννοια αυτή η πιο σημαντική του συμβολή είναι να βοηθούν τους καλλιεργητές να διατηρούν την ποσότητα του άνθρακα που δεσμεύεται στα γεωργικά ιστορικά εδάφη, αλλά τα μέτρα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην, ε, επίσης και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Τα αγροπεριβαλλοντικά και τα σοκομικά μέτρα αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός μηχανισμός ενθάρρυνσης αποθήκευσης του άνθρακα στα εδάφη και της ε, ε, φυτικής κάλυψης στην Αγγλία. Και υπάρχει ένα δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στην Αγγλία όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άμβληση της κλιματικής μεταλλαγής της κλιματικής αλλαγής συγγνώμη, είναι μόνο ένα από τα δημόσια αγαθά ε, στα οποία ο πυλώνας 2 της ΚΑΠ δραματίζει ζωτικό ρόλο και ίσως θα θέλατε να μάθετε ότι ο οργανισμός μας τελευταία δημοσίευσε κάποιες έρευνες που αξιολογούν τις συνολικές ανάγκες μιας ε, διαχείρισης περιβαλλοντικών ε, γεών στην Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, μια σημαντική προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε μια συνέχεια σε όλα αυτά τα μοντέλα. Τα μέτρα αυτά δεν θα είναι ποτέ ο βασικό μηχανισμό βελτίωση ενεργειακή αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία ή στη μείωση των αερίων εκπομπών θερμοκηπίου ε, μεθανίου και πρωτοξιδίου του αζότου από την παραγωγή, αλλά μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε ορισμένες σημαντικές εξοικονομήσεις ως υποπροϊόντα μιας διαχείρισης που είναι σημαντική για άλλους λόγους. Ούτε είναι οι βασικοί μηχανισμοί για την ενθάρρυνση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από βιοκαύσιμα ή βιομάζα. Ωστόσο, ενθαρρύνοντας την παραγωγή ε, καυσίμων από τα δάση, μπορούν να αντικαταστήσουν την παραγωγή από ενεργειακές ε, καλλιέργειες και μάλιστα κατά τρόπο που να βοηθήσουν στην άμβληση της κλιματική αλλαγή και να υποστηρίξουν τη βιοπικιλότητα. Ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό ε, σημείο ή στοιχείο της αγροπεριβαλλοντικής προσέγγισης για ε, η εξοικονόμηση του άνθρακα είναι συνεπής με τις βασικές αρχές της βιωσιμότητας. Οι, αυτές, η εξοικονόμηση αυτή του άνθρακα προκύπτει από μια διαχείριση η οποία επίσης ε, στηρίζει την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, ε, διαφυλάσσει την ε, βιοπικιλότητα και βοηθάει στην διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου. Όλα αυτά τα μέτρα είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στην άμβληση των κλιματικών μεταβολών. Ε, Βεβαίω όλα αυτά σχετίζονται και με την ε, παραγωγή τροφίμων. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε μια 20ετή εμπειρία ε, ολοκληρωμένων αγροπευρελοντικών μέτρων σε σχέση με την γεωργική παραγωγή και σε, όλα, όλους, σχέση με όλους τους τύπους καλλιέργειας. Και η εμπειρία μου δείχνει ότι θα πρέπει να προβούμε σε ένα πολύ προσεκτικό σχεδιασμό σεβόμενοι το περιβάλλον. Εδώ κλείνει η ομιλία μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι βρήκαν τις παρουσιάσεις αυτές πολύ ενδιαφέρουσες και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα την πρώτη συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά. Ο εισηγητής από την Επίτροπη Ήτρε θα πάρει το λόγο. Η Επιτροπή εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές, τον εισηγητή μάλλον, για την εξαιρετική του δουλειά. Και θα ήθελα να προσθέσω κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες στα πλαίσια της ε, δική μας προοπτικής μας φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες. Καταρχάς θα πρέπει νομίζω να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει περισσότερα μέσα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες κατά από τις οποίες γίνεται η επαφή ανάμεσα στο κλίμα και την παραγωγή. Βιοκαύσιμα, ένα θέμα. Πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Λιπάσματα, λιπάσματα όμως οικολογικά, αηφόρα, όπως επίσης και εκμετάλλευση όλων των αποβλήτων τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια της γεωργικής εκτινοτροφικής δραστηριότητας. Μία πιο έντονη και πιο αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα και σε τομείς όπως ε, η πληροφορική θα ε, βοηθήσει να βελτιώσουμε τους τρόπους παραγωγής και να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα μέσα παραγωγής τα οποία έχουμε και να μειώσουμε κατά συνέπεια ε, τα αέρια του θερμοκηπίου και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Ως προς αυτό τον τομέα λοιπόν εμείς ενδιαφερόμεθα είναι εξαιρετική η δουλειά την οποία ακούσαμε πάντως μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Μαγκίνες, η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για τις παρουσιάσεις τους. Έχω δύο ερωτήσεις να θέσω. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η κατάσταση του εδάφους. Σαν εμπειρογνώμονες μπορείτε να μας παρουσιάσετε μια η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τις οποίες εσείς προκρίνετε. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά που μας είπατε έχουν σημασία αλλά καλύπτεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ε, χώρο και εφόσον τα θέματα τα κλιματολογικά είναι αυτή τη στιγμή κατεπήγοντα και οξυμένα ποιες είναι οι προοπτικές ε, τις οποίες έχουμε, μία, δύο, τρεις προοπτικές πάνω σε αυτές να βασίσουμε την προσπάθειά μας. Ε, άκουσα από τον Φρανκο Μάρα κάποια αποτελέσματα σχετικά θετικά αν και περιορισμένα θα έλεγα, στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών μεθανίου. Άκουσα μια ειλικρίνεια λοιπόν από πλευράς του και αυτό με χαροποίησε, γιατί δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό από τους εμπειρογνώμονες να παραδέχονται τους περιορισμούς τους. Από την άλλη είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι πιστώσεις τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας για την καλύτερη διακίνηση και αλληλοεπικοινωνία των γεωργών σχετικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούν. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τα αποτελέσματα της έρευνας και με την εφαρμογή αυτών των αποτελεσμάτων. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συμπληρώσουμε τα κενά τα οποία έχουμε αναμφισβήτητα. Και σε σχέση με ε, την έννοια του δημοσίου αγαθού, τι εννοώ εδώ. είναι βασικό χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Βέβαια ποσοτικά δεν είναι προσμετρήσιμο. Εσείς πιστεύετε ότι εμείς σαν εμπειρογνώμονες ή σαν άνθρωποι που λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, τους γεωργούς να χρησιμοποιούν τα μέσα τα οποία προτείνεται σε αυτή τη φάση ή είναι πρόωρο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ και εγώ τους τρεις ε, εισηγητές. Ο... Η έκθεση Λεφόλ επίσης είναι εξαιρετική και νομίζω ότι θα συζητηθεί, πρέπει να συζητηθεί όπως της αξίζει αργότερα. Οι ερωτήσεις μου έχουν σχέση με τις ερωτήσεις της κυρίας Μαγκίνες. Μία διευκρίνηση, αν γίνεται, ε, ό,τι αφορά την προέλευση του πρωτοξιδίου του αζότου και ποια είναι η, ποιο είναι το εύρος της κτηνοτροφίας και πώς έχουν αλλάξει τα μεγέθη. Ε, και σε σχέση με τις ανάγκες ε, ε, σε κτηνοτροφικά είδη. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες διευκρινήσεις εδώ. Επανέρχομαι στις συζητήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της γεωργίας και της αύξησης της οικονομικής της αποδοτικότητας. Τι πιθανές λύσεις έχουμε. Η ερώτηση που θέλω να κάνω σχετικά είναι ποια είναι τα μεγάλα κέρδη σε σχέση ε, με την ε, διαχείριση ε, κτηνοτροφικών καλλιεργειών σε σχέση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες γιατί είναι δύο χωριστά θέματα. Επίσης η διαχείριση χαρτολιβαδικών εκτάσεων ε, ε, ειδών που μοιάζουν με το τριφύλι, ποικιλίε ε, τριφυλιού κλπ. Τώρα για το μεθάνιο ένα βασικό μήνυμα είναι καλύτεροι συντελεστέ μετατροπή. Αυτούς τους χρησιμοποιήσαμε εδώ και πολλά χρόνια για την βιομηχανία των τροφίμων. Επίσης ε, διαχείριση κοπριάς, ε, ιδαρούς λάσπης ε, και αυτό είναι σημαντικό για να δούμε πού πρέπει να επικεντρωθούμε και να επιτύχουμε τα περισσότερα ωφέλη. Για το πρωτοξίδιο του αζότου η μείωση αυτή καθ' αυτή είναι που πρέπει να μετράμε και είναι καθοριστική παράμετρος, υπάρχουν και άλλοι δείκτες. Δηλαδή πού είναι πιο εύκολο να επιτύχουμε στην πρώτη πενταετία τα μεγαλύτερα ωφέλη, γιατί είναι σημαντικό αυτό σε σχέση με τα ρύθμιση και τις προτεραιότητες της ΚΑΠ στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Λάιον. Ο κύριος Χάρσλινγκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους εισηγητές και τον ε, τους, ε, τον εισηγητή τον κύριο Λεφόλ. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς τους δύο τελευταίους ομιλητές ε, για τις εκπομπές ε, λέμε ότι είναι κάτω από το 10% επίσης εισαγωγές ζωοτροφών ε, σημαίνουν εκπομπές σε άλλες χώρες ε, από ε, εισαγωγές από την Αργεντινή, τη Βραζιλία κλπ. Αυτά που παρουσιάζονται στο ισοζύγιο του κλίματος νομίζω ότι και αυτά πρέπει να τα προσμετρήσουμε γιατί ενδεχομένως διπλασιάζουν τα ποσοστά αν λάβουμε υπόψη μας και τις εκπομπές ε, και τις περιβαλλοντικές ζημίες σε χώρες όπως Βραζιλία και Αργεντινή. Δεν πρέπει λοιπόν αν είμαστε τίμοι να τα συμπεριλάβουμε στους ισολογισμούς μας και ε, στα ισοζύγια. Τώρα, η διατροφή, η αποτελεσματικότητα τροφίμων, ε, προσφοράς ε, ε, τροφίμων ε, και διατροφή των ζώων. Οι αγελάδες δεν παίρνουν αποκλειστικά χόρτο, άρα ανατρέπονται και εδώ κάποια ισοζύγια αν κάνουμε ειλικρινείς υπολογισμούς γιατί έχουμε άλλους συντελεστές. Η διατροφή των ζώων είναι πιο εντατική με δημητριακά και όχι μόνο με χόρτο. Η προστασία της Γρελανδίας είναι πολύ σημαντική επίσης σε σχέση με την προστασία του κλίματος. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, ε, εδάφη όπου καλλιεργείται χόρτο. Ε, επίσης η αποθήκευση του ε, άνθρακα ε, σε, στο έδαφος. Ε, θα πρέπει να δούμε τι δυναμικό ε, υπάρχει γενικότερα. Τώρα, τα διαφορετικά συστήματα χρήσης της γης, η βιολογική γεωργία είναι αποτελεσματικότερη σε σχέση με την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι κάτι δηλαδή που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας παράλληλα με άλλα μέτρα. Και τέλος, η παραγωγή βιοαερίου ε, κατά πόσον συμβάλλει στην αύξηση ε, της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. În χωρίς μικρόφωνο. Μ' ακούτε τώρα. Πήγα το 95-96 στο Πανεπιστήμιο ή στα Αγγλία για να ακούσω μία ομιλία για την παγκόσμια ε, θέρμανση ε, και μας έδωσαν και ορισμένα στοιχεία ε, μέσα σε 30 χρόνια. Από τότε δεν άλλαξαν πολλά. Συνεχίστηκε και η αύξηση της θερμοκρασίας και άλλαξα και τις καλλιέργειές μου. Άρχισα λοιπόν να παράγω σκληρό σύτο γιατί μας είπαν ότι ε, το κλίμα της Αγγλίας θα γίνει όπως είναι τώρα της Ισπανίας. Οπότε θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε σκληρό σίτο και άλλοι όχι μόνο εγώ. Όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα γιατί είχαμε παγετό καθυστερημένα στην εσοδεία για 11-12 χρόνια το πάλεψα το πράγμα και πρόσφατα μας έδωσαν κάποιες προβλέψεις ε, τον Αύγουστο του 2008 για ήπιο χειμώνα ε, σε σχέση με την παγκόσμια υπερθέρμανση. Οπότε ε, προσαρμόστηκα κι εγώ σε σχέση με τη, την οτροφία μου. δεν συνέβη αυτό. Επίσης ε, υπάρχουν ε, ε, μετεωρολογικές προβλέψεις οι οποίες στηρίζονται, ανέφεραν αυξημένη ηλιοφάνεια που έπεσαν περισσότερο μέσα. Το μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει θερμοκήπια και το διοξίδιο του άνθρακα εκεί για την καλύτερη και γρηγορότερη αύξηση των φυτών. Επίσης, ο ε, ο δόκτωρ ε, ε, καθηγητής Φράνκο Μάρα είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό των των αερίων του θερμοκηπίου. Έχουμε μετρήσει όμως που δείχνουν άπειρο ελάχιστες ποσότητες. Ε, αναφέρομαι επίσης ποσοστά που προέρχονται από μυρικαστικά ή από βακτήρια. Θα πρέπει να τα διαφοροποιήσουμε και τα μυρικαστικά και αγρία ζώα φαίνεται να ε, ε, έχουν να είναι περιορισμένη η πηγή. Ε, το, η πάντοτε βεβαίως παρήγαγε μεθάνιο. Πού υπάρχει διαφοροποίηση τώρα. Ε, βεβαίως όχι να οργώνομαι παραδοσιακά ε, χορτολιβαδικές, παραδοσιακές χορτολιβαδικές εκτάσεις όμως τώρα ε, βλέπουμε ε, να έχουμε εντατικοποίηση στις αρωτρές ε, καλλιέργειες και οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα αυτές τις ομιλίες με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που θεωρώ ότι αποσιάζει από αυτή τη συζήτηση είναι μια συνολική αξιολόγηση της γεωργίας. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι η μόνη μέθοδος, η μόνη μέθοδος για τη δέσμευση του άνθρακα είναι η φωτοσύνθεση. Και στη φωτοσύνθεση η γεωργία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε πόσες εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο ε, καλλιεργούνται από τη γεωργία, αρδεύονται ε, ε, εκτάσεις όπου είναι μικρότερη η δυνατότητα απαγίδευσης του άνθρακα. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποιοι σχετικοί υπολογισμοί. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι βλέπουμε τα πράγματα όχι σφαιρικά. Στο Κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε μια διοργάνωση με τον τίτλο «Λιγότερο κρέας, λιγότερη θερμότητα». Στο Time πριν από δύο ε, εβδομάδες έγραφε «Σώσε τον πλανήτη να τρώτε περισσότερο βοδινό κρέας». Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα και παρόλο που διευκρινίστηκαν κάποια πράγματα εδώ σήμερα το πρωί, δηλαδή πρόκειται και για τις δύο αυτές ε, στάσεις, δηλαδή από το, το πώς εκτρέφονται τα ζώα από τη μία, και εδώ θα πρέπει να πούμε στην κοινή γνώμη ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Δηλαδή ότι υπάρχει και παραγωγή κρέατος η οποία δεν είναι επιζήμια όσον αφορά την κλιματική μεταβολή. Αντίθετα μπορεί να οδηγήσει ή να συμβάλλει στην παγίδευση του άνθρακα και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Θεωρώ ότι η έκθεση του συναδέλφου Λεφόλ είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσο δεν πρόκειται για μια ευκαιρία για τη γεωργία και για μας τους πολιτικούς να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές μεταβολές, γιατί πρόκειται εδώ για ένα δημόσιο αγαθό είναι αυτή μια δυνατότητα να δικαιολογήσουμε τις πληρωμές στην γεωργική πολιτική. Τι μέτρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε με το κρασί, ε, με τις συνοκαλλιέργειες που βρίσκονται σε ευθύνουσα κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκεί όπου τα έδαφος είναι επικλινές. Δεν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στην πολιτική γεωργίας να υιοθετηθούν νέα μέτρα. Are cuvântul euh. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν, κ. Μποβε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί πιστεύω ότι το γεγονό ότι έθεσε αυτό το θέμα επιτάπητος είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω του παρεμβαίνοντες γιατί ε, έριξαν φω στη συζήτηση. Και δεν ξέρω, παίρνω στο λόγο, αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω. Γιατί έχω την εντύπωση ότι περπατάμε ανάποδα. Με... Κανείς δεν μίλησε για την ευθύνη μιας κοινή γεωργικής πολιτικής στην παρούσα συγκυρία. Γιατί 30 έτη κοινή γεωργικής πολιτικής κατασκεύασαν ένα μοντέλο ανάπτυξης παραγωγιστικό που μας οδήγησε σε αδιέξοδο. Σήμερα γίνεται με πιστή μονικοφανή τρόπο λόγος για τις επιπτώσεις αυτού του μοντέλου. Θεωρώ ότι αυτό είναι παράδοξο και μας εξηγούν ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ψηθούμε στους επιστήμονες για να μας εξηγήσουν ότι οι αγελάδες ε, τρώνε χόρτο. Ε, δηλαδή όλα στοιχεία της αγρονομίας, βασικά στοιχεία της αγρονομίας που γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά εδώ και 30 χρόνια χρηματοδοτήσαμε τους ε, καλλιεργητές για να κάνουν το αντίθετο. Και όταν ε, δίναμε ένα γαλλικό φράγκο εδώ και πολλά χρόνια, 3 εκατομμύρια φράγκα για να αρδεύεται ένα ε, χωράφι με καλαμπόκι, δίναν 300 φράγκα για ένα εκτάριο χορτολιβαδικό. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά παράδοξα. Τώρα, μιλάμε για την εκτροφή. Ε, όπως είπε ο κύριος Χόσλινγκ, αναφέρθηκε στις εισαγωγές. Οι εισαγωγές ε, σόγιας, 22 εκατομμύρια εκτάρια από την Λατινική Αμερική, που θα πρέπει να ενταχθούν στον, του, στον Ευρωπαϊκό Ισολογισμό του Άνθρακα. Και όχι ε, της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε αυτή την ευθύνη γιατί κάνουμε αυτές τις εισαγωγές και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα ένα άλλο στοιχείο. Αναπτύξαμε επιστημονική έρευνα σε ένα ιδιαίτερο μοντέλο μοντέλο παραγωγιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή όσο πιο ε, πολλοί παράγοντε, όσο περισσότερο υποστηρίζουμε την παραγωγή. Τώρα, τι γίνεται με του σπόρου. Κανεί δεν μίλησε για του σπόρου. Το αγρονομικό μοντέλο των σπόρων σήμερα είναι πρωτίστω καταναλωτικό των λιπασμάτων. Και για να λειτουργούν αυτοί οι σπόροι χρειάζονται πάρα πολλά λιπάσματα. Αυξάνεται λοιπόν συνεχώ η χρήση λιπασμάτων. Και όλες οι έρευνες που πηγαίνουν προς μια άλλη κατεύθυνση Προφανώς σήμερα δεν το στηρίζει κανείς. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε να αμφιβόλω ένα μοντέλο το οποίο επιβάλλεται σήμερα από τις μεγάλες εταιρείες που παράγουν αυτά τα λοιπάσματα. Γιατί υπάρχει μια ξεκάθαρη διασύνδεση σήμερα και όλοι το γνωρίζουμε, θα μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες, μεταξύ των αγροχημικών ε, βιομηχανιών και αυτών των ε, καλλιεργιών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε αυτό το μοντέλο, μην έχουμε φόβο να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο. Μας λένε ότι θα πρέπει να εντάξουμε την κοπριά στο έδαφος, να μην την διαχέουμε πάνω από το έδαφος, να την βάλουμε μέσα στο έδαφος. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να μην ε, την παράγουμε, γιατί τον εκτρέφουμε ζώα πάνω στο πετόν και στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε αυτήν την υγρή κοπριά, νομίζω ότι είναι τελείως ηλίθιο. Ε, το καλύτερο να κάνουμε κομπριά, να κάνουμε κομποστοποίηση, να δεσμεύουμε τον άνθρακα και στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε αυτή την κοπριά. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, δώσουμε αυτό το μοντέλο, πρέπει να ξεφύγουμε αυτό το μοντέλο. Και νομίζω ότι έχει, θα πρέπει να πούμε για την έκθεση του Στεφάν Λεφόλ, Εάν θεωρήσουμε σήμερα ότι αυτό το θέμα είναι κεντρική σημασία, χρειαζόμαστε μια νέα κοινή πολιτική γεωργίας που γυρίζει την πλάτη σε 30 χρόνια ολοσχερούς ε, καταστροφής από διάφορες της ε, γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Ε, ευχαριστώ πολύ και τους επιστήμονες. Έχω γράψει εδώ τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, κατάλαβα ότι εδώ δεν υπάρχουν απλές ε, λύσεις και δεν είναι δυνατόν να σκέφτεται κανείς με κλισέ, στερεότυπα. Η μη χρήση δεν είναι εν γέννη θετική. Δηλαδή λέγεται συνήθως ότι έχει εγκαταληφθεί η γεωργία, δεν υπάρχει χρυσή και αυτό δεν είναι καλό για το διοξείδιο του άνθρακα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε από ένα εντατικό αγαθό ένα εντατικό κακό. Έγραψα η εντατική γεωργία είναι καλή κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη ερώτηση προς τους επιστήμονες είναι τι είδους γεωργία θα μας συστήνατε. Το πρόβλημα τα προβλήματα στην ε, πολιτική χρειάζονται απλές, απλουστατιστικές απαντήσεις για να μπορεί να μας καταλαβαίνει και ο λαός. Πάντοτε είναι αυτό το θέμα επικοινωνία με του πολίτε. Δεύτερο πρόβλημα. Συμφωνείτε ότι η Γεωργία δεν είναι το πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε ή θα πρέπει να αποτελέσει τη λύση του προβλήματος. Αληθεύει αυτό. Εγώ ίδιος είμαι Γεωργός και αυτή είναι η θα πρεπει να αποτελεσει τη λυση του προβληματο αληθευει αυτο εγω ιδιο ειμαι γεωργο και αυτη ειναι η ελπιδα που έχω για το μέλλον, να μπορούμε και εμεί να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματο. Και το τρίτο ερώτημα το έθεσε ήδη η συνάδελφο Μαγκίνες. Ποιες είναι οι προτεραιότητε που προτείνετε εσεί για τη Γεωργία Δηλαδή, πού βρίσκεται το δυναμικό αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ τους επιστήμονες για τις ομιλίες τους. Ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο κύριο Λεφόλ που εκτιμώ πολύ και που έκανε μια σωστή διαπίστωση δηλαδή οικονομική διαχείριση των πόρων, γιατί είναι πεπερασμένη. Ε, όμως επιφυλακτικά αντιμετωπίζω την ιστερία σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα. Πριν από 25 χρόνια ε, ίδρυσα έναν σύλλογο για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, για τη διατήρηση των πεπερασμένων πόρων. τώρα ε, θα πρέπει να δω αν είναι σοβαρά τα στοιχεία που ε, δίνουν οι επιστήμονες για το διοξίδιο του άνθρακα τελευταία όλο και περισσότερες ε, αναφορές με τους εξής τίτλους για παράδειγμα προβάλλονται στον τύπο που αφορούν τους τα κλιματολογικά δεδομένα, ε, την αλλαγή ε, κλίματος και τη σχέση τους με τη γεωργία, ε, το LPCC κλπ. Υπήρξαν επίσης και τηλεοπτικά προγράμματα που αναφέρεται σε, αναφο... σε ψευδή δεδομένα Πώς θα συνεχίσουμε την έρευνα λοιπόν με βάση ψευδή δεδομένα. Βεβαίως είμαι πολιτικός πολλά χρόνια ε, για να δέχομαι τα πάντα ως ειλικρινή. Το 80-81 ε, γίνονταν προβλέψεις σε σχέση με την επόμενη 20 ετία και από Γερμανούς επιστήμονες ή από ε, Βρετανούς που ανέφεραν ε, εξέλιξη ε, με διαφορετικά είδη καλλιεργιών. Ε, το όλο και περισσότερο ε, βλέπουμε ιστερικές αντιδράσεις και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι υποπτεύεστε κι εσείς ότι ενδεχομένως πίσω από όλα αυτά κρύβονται οικονομικά συμφέροντα. έχω και μετεωρολογικό ε, δελτίο το οποίο παρακολουθώ και ε, έχω ε, δυνατότητα από το 89 να έχω μετρήσει της θερμοκρασίας κάθε 10 λεπτά. Στη δική μου επιχείρηση η μέση θερμοκρασία ε, έξω στους αγρούς ήταν 9,14 βαθμοί. Η μέση αυτή θερμοκρασία δεν ε, έχει ε, παρατηρεί διαφορές και αυξήσεις θερμοκρασίας δεν έχουν παρατηρηθεί. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αυξάνεται η θερμοκρασία ε, όπως αναφέρεται ενώ στη δική μου ε, έκταση ε, δεν παρατηρείται. Βλέπω ότι δεν είναι πάντοτε 100% αξιόπιστα τα επιστημονικά δεδομένα. Μήπως λοιπόν στηρίζονται περισσότερο σε αστρολογικά δεδομένα παρά μετεωρολογικά. Ε, δεν νομίζω ότι ε, υπάρχουν τόσο μεγάλες ε, διαφορές και βέβαια από πολλούς δεν λαμβάνονται και σοβαρά. Επίσης, αν το διοξείδιο του άνθρακα επηρεάζει το κλίμα, γιατί στη Βαβαρία διαπιστώνεται το εξής, αξιόπιστα. Το 1971, ήπιος χειμώνας ε, μετά το 85 πάλι ήπιος η χειμώνας ε, το Μάιο, τον Αύγουστο δεδομένα για την, ε, τις καλλιέργειες, ε, ε, αμπελοκαλλιέργειες κλπ. Ε, αναφορές σε σχέση με τα οποροφόρα. πάλι τα επόμενα χρόνια ε, ήπιος σε κεράσια το Μάρτιο, ε, τα οποία δεν εισήχθησαν ε, αεροπορικός από την Νότια Αμερική. παλιότερα λοιπόν αυτές είναι αναφορές από προηγούμενα έτη. Αν ήταν τόσο ήπιοι οι χειμώνες και τότε, δεν μπορεί να φταίει το, η εντατική κτηνοτροφία και η αύξηση στην ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα. άρα λοιπόν, πού είναι τα αξιόπιστα δεδομένα και η πραγματική εξέλιξη στο κλίμα. Ευχαριστώ κύριε Ντές. Θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί ε, Ευρωπαίοι συμμερίζονται το σκεπτικισμό σας και αυτό έχει άμεση σχέση με τον ρόλο τον οποίο παίζουν οι εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να μιλήσουν πιο ξεκάθαρα. Και οι πολιτικοί παίζουν κάποιο ρόλο βέβαια επίσης γιατί θα πρέπει να είναι ρεαλιστές απέναντι στα θέματα των κλιματολογικών αλλαγών κύριος Βορτσιακόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι μάλλον συμφωνώ με τα σχόλια τα οποία έκανε ο κύριος Ντες. Αν δει ποια είναι η κατάσταση στην Πολωνία φέτος, ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα σκληρός, είναι ιδιαίτερα σκληρός και όταν βλέπει ε, κανείς να επικρατούν τέτοιες θερμοκρασίες διαρωτάται ε, αν πράγματι υπάρχει θέμα ε, αύξησης της θερμοκρασίας. Μετά από τις τρεις παρουσιάσεις τις οποίες άκουσα σήμερα, εγώ ανανεώνω την εμπιστοσύνη την οποία έχω απέναντι στην έρευνα και στους ερευνητές και τα στοιχεία που μας δίνουν. Υπάρχουν όμως ε, κάποιες αποστάσεις τελικά ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι κάνουν την έρευνα και ανακοινώνουν τα αποτελέσματά της και σε αυτούς οι οποίοι καλούνται ή και δεν καλούνται μερικές φορές να την εφαρμόσουν, να τα εφαρμόσουν τα αποτελέσματα αυτά. Έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατηγορία, τους γεωργούς. Οι γεωργοί έχουν μια αντίληψη για τα πράγματα. Όταν λέμε στους γεωργούς λόγια μεγάλα σχετικά με τις επιπτώσεις τις οποίες έχουν ε, τα ζώα τα οποία εκτρέφουν στο κλίμα, δημιουργούμε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να βελτιωθεί. Περιμένουν απαντήσεις οι γεωργοί και στοιχεία και λεπτομέρειες τις οποίες προς το παρόν ακόμα δεν έχουν πάρει. Πρέπει η επιστημονική πληροφορία να μεταφερθεί σαν μήνυμα προς τους γεωργούς οι οποίοι εφόσον πιστούν θα προσπαθήσουν να αντιθέσουν σε λειτουργία. Όλοι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια για να πείσουμε τους γεωργούς με τον σωστό τρόπο. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες έχουν άλλοι δύο συνάδελφοι ζητήσει το λόγο ο κύριος Καπούλα Σάντος πρώτος. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις εξωτερικές παρουσιάσεις, να ευχαριστήσω και τον κύριο Λεφόλ. Νομίζω ότι η έκθεσή του είναι ιδιαίτερα συνεκτική. Τοποθετεί το θέμα της κλωματολογικής αλλαγής στο σωστό πλαίσιο και επιτρέπει έτσι να ξεκινήσει η συζήτηση την οποία όλοι χρειαζόμαστε για το μέλλον της ΚΑΠ δεν παρέχει μόνο διαγνωστικά μέσα, αλλά κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε εφαρμόσιμα πολιτικά βέβαια μέτρα. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες καταρχάς ακούσαμε μία ολόκληρη σειρά προτάσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να καταπολεμηθεί το πρόβλημα. Ιδανικά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς τα μέσα αυτά από κοινού. Βέβαια το κόστος θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Βασικά λοιπόν ποια είναι η καλύτερη σχέση στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, για το κόστος ε, σαν παράδειγμα η αναδάσωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι αποτελεσματικό μέσο. Οικονομικά είναι αποδοτικό μέσο, βραχυπρόθεσμα μάλιστα. Έχω επίσης μία ερώτηση προς τον εισηγητή. Αναφέρθηκε και ο εισηγητής στα της αναδάσωσης. Αλλά δεν τόλμησες, και συγγνώμη που το θέτω έτσι άμεσα, να κάνεις ένα βήμα επιπλέον να πεις ότι απαιτείται μια κοινή πολιτική για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες μέχρι τώρα για την απόκτηση μιας κοινή πολιτικής απέτυχαν. Αν θέλουμε να συγκρατήσουμε τον άνθρακα εντός του εδάφους, πρέπει να βάλουμε στόχους κοινού στον τομέα των δασών σαν ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ερωτών Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Εδώ και χρόνια ακούμε αποκαλυπτικούς τίτλους και καταστροφολογίες σε σχέση με το θέμα αυτό. Εγώ όταν σπούδασα στο Πανεπιστήμιο σπούδασα ε, σχέσεις ε, και έκανα μελέτες για το κλίμα Ήδη υπήρχαν έρευνες για την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά θερμή υπερθέρμανση του πλανήτη υπήρχε και παλιότερα, ακόμα και την εποχή των δεινοσαύρων. Συνεπώς δεν μιλούμε για κάτι καινούριο, αλλά κάτι που έρχεται από την αρχαιότητα. Είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας, η, συγγνώμη, λέει, μιλήτρια η ιστορία του πλανήτη. Γι' αυτό με κατέπληξε όταν ε, άρχισαν, ε, να μιλάτε, ε, να γίνεται λόγος για φαινόμενα αποκάλυψης. Ε, ότι θα, άλλαζε, θα αλλάξει ριζικά η μορφή του πλανήτη. Όλα αυτά τα πράγματα μας ε, οδήγησαν στο να ακούμε και να διαβάζουμε αυτό που μας ε, αφηγούνται οι άλλοι και μας απειλούν. Και όλα αυτά με οδηγούν στην εξή σκέψη. Το κλίμα έχει δυναμικό χαρακτήρα, μεταβάλλεται. Ε, αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής ε, στην ιστορία, αλλά δεν πρόκειται να διχειούμε στην ε, υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό το νομίζω ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν πρόκειται να γίνουμε μάρτυρες αυτών των φαινομένων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης και είναι ένα θέμα το οποίο δεν σχετίζεται κατά κανένα τρόπο με έναν κλιματικό κατακλυσμό αλλά είναι ένα θέμα ηθικής ευθύνης, ηθικού χρέους ως ανθρώπινα όντα, να σεβόμεθα το περιβάλλον στο οποίο ζούμε για να είναι πιο ευχάριστο για μας και για τα παιδιά μας. Ωστόσο, δεν δέχομαι ε, κάποιοι που στρέφονται κατά της ε, γεωργίας να εκμεταλλεύονται αυτό το θέμα και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να δεχόμαστε τον εμπλουτισμό πολλών ε, προσώπων και κάποιων άλλων που κερδίζουν βραβεία Νόμπελ με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει πληρώσει το τίμημα για την βλάβη που έκαναν στην ανθρωπότητα αυτά τα, αυτοί οι άνθρωποι. Ε, και έχει γίνει εκμετάλλευση και πολλών φυτογειονομικών θεμάτων από μεγάλες επιχειρήσεις κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Ε, θεωρώ ότι όπως σας είπα πάρα πολλοί βασίστηκαν στην άγνοια Τρίτον, για να εμπλουτίσουν και να αποφεληθούν οι ίδιοι. Για μένα η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να μας βοηθήσει τους ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για μας και τους απαγόνους μας. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να στραφεί ο δεύτερος πυλώνας στην ανάπτυξη της γεωργίας. Ε, και ο κύριος Λεφόλ αναφέρεται πολύ σωστά στην σωστή διαχείριση της δασοκομείας στην έκθεσή του. Ε, θα πρέπει αυτός ο πρωτογενής τομέας να συνεχίσει να διατηρεί τη θέση του. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, διάβρωση του εδάφους και την, να καταπολεμήσουμε και τα φαινόμενα προδοσίας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Η κοινή γεωργική πολιτική του μέλλοντος θα πρέπει να είναι μια ισχυρή πολιτική γεωργίας όπως ήταν στο παρελθόν με την έκθεση του συγητού. Έχω μόνο μία αμφιβολία ε, σε σχέση με το αποτύπωμα του άνθρακα με την επισήμανση του αποτυπώματος του άνθρακα. Αν δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική μέθοδος για την αξιολόγηση του αποτυπώματος του άνθρακα, ας μην ε, διακινδυνεύσουμε να κάνουμε κάτι που είναι ολιστηρό έδαφος, που ολιστηρό έδαφος. Εάν δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος, ε, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα αυτά είναι ασφαλή και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς ότι οι υπόλοιπε τρίτε χώρε πρόκειται να αναλάβουν επίση τα, εγκεκριμένα, τα ενδεδειγμένα μέτρα. Θα υποχρεώνουμε του καλλιεργητέ μα να καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια χωρί να έχουμε την αμοιβαιότητα των άλλων. Εάν δεν έχουμε λοιπόν μια επαρκή επιστημονική βάση, να μην ε, το πράξουμε, να μπούμε σε αυτό το χωράφι. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Ο επόμενος θα ακολουθήσει αφόκους με τους υπόλοιπους τρεις ομιλητές. Δίνω και πάλι το λόγο στους εμπειρογνώμονες για να σχολιάσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Τους παρακαλώ να τηρήσουν ένα χρονικό όριο, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ακρόαση έγκαιρα. Κύριε Ρεκόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θέλω να μιλήσω σε σχέση με τη γεωργία και τις τεχνικές διατήρησης. Όλοι χρειαζόμαστε τρία γεύματα τη μέρα και στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, είναι τυχεροί αν έχουν ένα γεύμα τη μέρα. Η γεωργία έχει να παίξει τεράστιο ρόλο στην εξασφάλιση τροφίμων, ινών στις κοινωνίες μας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα εδάφους που διαταράσσεται από τα γεωργικά συστήματα. Η εντατική άρρωση οδηγεί σε διάβρωση και σε άλλες μορφές υποβάθμισης. Με αυξανόμενη ένταση άρρωσης ε, ε, με, μειώνοντας την ένταση της ε, έντασης με άλλα συστήματα ε, ε, σποράς ε, μπορούμε να έχουμε πολλά ωφέλη μειώνοντας και βραχυπρόθεσμα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οι αγρότες εδώ καταλαβαίνουν ότι αν μειωθεί το όργωμα τότε διαταράσσεται λιγότερο το έδαφος και μειώνεται η ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται. Ε, μειώνονται επίσης και τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται για το όργωμα. Μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε την ένταση της ε, ε έτσι μπορεί να δεσμευτεί και το διοξίδιο του άνθρακα από την φωτοσύνθεση. Οι διαχειριστές γεωργοί έχουν ε, σημαντικό ρόλο να παίξουν εδώ. Είναι σημαντικό να έχουμε επιφάνειες πρασίνου που θα δεσμεύουν ε, το διοξίδιο του άνθρακα όσο γίνεται περισσότερο για τη διατήρηση των συστημάτων παραγωγής μας. Συνοψίζω, ε, ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στη Γεωργία είναι να ελαχιστοποιήσουμε την διατάραξη του εδάφους, γιατί η έκκληση του διοξιδίου του άνθρακα είναι αναλογικό προς τη διατάραξη αυτή των εδαφών. Επίσης, τα συστήματα των καλλιεργών μπορούν να αλλάξουν, συστήματα αμυψής σποράς που θα αποσκοπούν σε ε, διατήρηση επιφανειών πρασίνου. Έτσι μπορούμε να έχουμε πρόοδο και να μειώσουμε τον, αντίκτυπο, τον επιζήμιο αντίκτυπο της γεωργίας στο κλίμα. σταματώ για να προλάβουν και οι άλλοι να απαντήσουν. Ο Φρανκ Ομάρα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν τη δική μου παρουσίαση. Πρώτον, ποιος είναι ο ρόλος της γεωργίας σαν τμήμα του προβλήματος και τμήμα της λύσης του πρόβληματος. Κάποιοι από τους ομιλητές αμφισβήτησαν την συνεισφορά της γεωργίας στη δημιουργία του προβλήματος. Είναι αλήθεια αυτό. Τα ζώα πάντα υπήρχαν. Οι κλιματολογικές αλλαγές είναι σχετικά πρόσφατο θέμα και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα ακριβώς του τρόπου με τον οποίο καταλογίζονται αν θέλετε οι προσπάθειες, οι ευθύνες μάλλον και οι προσπάθειες κατανομής των ευθυνών στη Γεωργία. Αν πάρετε μια χώρα σαν τη Γεωργία, σαν την Ιρλανδία συγγνώμη, βλέπετε ότι συνολικά οι εκπομπές της χώρας από το 90 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 22%. Οι εκπομπές συνολικά Παρ' όλα αυτά οι γεωργικές εκπομπές έχουν μειωθεί και η παραγωγή τροφίμων έχει αυξηθεί. Συνεπώς λοιπόν η γεωργία έχει παίξει πολύ μικρό ρόλο στην αύξηση των εκπομπών από το 1990 και ταυτόχρονα έχει δώσει τη δυνατότητα στην χώρα μου να έχει και περισσότερα τρόφιμα και να εξάγει και περισσότερα τρόφιμα. Είναι λοιπόν υπερβολικό να στοχεύεται η γεωργία σαν βασικό συνεισφορέας για την αύξηση των, των αερίων του ε, θερμοκηπίου και συμφωνώ με την άποψη αυτή. Αν δει κανεί λοιπόν ε, την Ιρλανδία και δει ακριβώ ε, από πού προέρχεται η αύξηση αυτή, οφείλεται κυρίως στην αυτοκίνηση τεράστια αύξηση των αυτοκινήτων και τεράστια αύξηση των χιλιομετρικών αποστάσεων που καλύπτουν τα αυτοκίνητα αυτά κατ' Και το σύστημα υπολογισμού το οποίο έχουμε και μέσα από το οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα υπολογίζει και την εκπομπή ε, αερίων από τη Γεωργία. Στην Ιρλανδία αντιπροσωπεύουν ε, το 25 με 30%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 19%. Ε, είναι σημαντικό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του συνόλου των εκπομπών τις οποίες παράγουμε ή προκαλούμε από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού αρχίζει και πού τελειώνει η ευθύνη της γεωργίας. Κάποιες άλλες ερωτήσεις αφορούν είναι η συνεισφορά των μυρικαστικών στην παραγωγή μεθανίου. Προέρχονται βέβαια εκπομπές και από άλλες πηγές όπως τα έλλη, κάποιες πηγές θερμές κτλ. Ε, βασική πηγή ε, βέβαια παραγωγής μεθανίου εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ε, τα μυρικαστικά. Αν ε, το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε και το οποίο έχει συμφωνηθεί λέγει κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι η εισαγωγή ζωοτροφών από άλλες χώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ίσως ε, να συνυπολογιστεί στην ε, παραγωγή αερίων από τις ε, γεωργικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν προσπαθούμε να στοχεύσουμε στον υπολογισμό του ενεργειακού ίχνους σε άνθρακα ή της ετικετοθεσίας η οποία αναφέρεται στην παραγωγή άνθρακα. Ε, και υπάρχει θέμα εδώ να δούμε πού θα ε, κατανείμουμε τις ευθύνε στη χώρα η οποία παράγει ή στη χώρα που θα κατανειμουμε την ευθυνε στη χωρα η οποια παραγει η στη χωρα που χρησιμοποιει το προϊόν. Όταν σαν παράδειγμα με ορυκτά καύσιμα οι εκπομπές συνυπολογίζονται σαν εκπομπές της χώρας που τα χρησιμοποιεί. Ενώ η παραγωγός χώρα όπως η Σαουδική Αραβία συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται. Ενώ όταν εμείς στην Ιρλανδία παράγουμε κρέας και το εξάγουμε σε άλλη χώρα χώρα, η Ιρλανδία, επιβαρύνεται από τις εκπομπές των αερίων τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτροφής. Αυτά είναι ενδιαφέροντα σημεία που θα απασχολήσουν και εσά τους πολιτικούς και εμάς τους εμπειρογνώμονες. Να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν πού είναι το καλύτερο μέρος για να παράγεται το τρόφιμο το οποίο έχει ανάγκη ο πλανήτης. Νομίζω ότι η βασική απάντηση λέγει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σπόρους που ε, ε, εισραίουν στην γεωργία για να μειώσουμε ε, την παραγωγή άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τις γέες που είναι διαθέσιμες και όχι να συμπεριλάβουμε νέες γέες στη γεωργική καλλιέργεια. Ίσως να μην το γνωρίζετε, δεν ξέρω ακριβώς τους αριθμούς, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ε, εξίσου ε, ίσες ποσότητες ε, εκπομπές ε, αερίου από τις νέες γέες οι οποίες εισάγονται σε χρήση κατέτος ε, με το σύνολο των εκπομπών από τις υπόλοιπες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Το θέμα λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε τα εδάφη που ήδη χρησιμοποιούμε με αποτελεσματικότερο τρόπο για την παραγωγή των τροφίμων μας ε, πριν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και νέες γέες. Όπως είπα λοιπόν στην ομιλία μου η Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι αρκετά αποτελεσματική σε σχέση με την ποσότητα των τροφίμων της, την οποία παράγει και σε σχέση με την παραγωγή εκπομπών κιλό τελικού προϊόντος το οποίο παράγει. Κάποιοι άλλοι ε, ομιλητές αναφέρθηκαν στην αποτελεσματικότητα παραγωγής τροφίμων. Το θέμα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα και για να σας διαβεβαιώσω θα ήθελα να πω ότι τα ζώα μας ε, ε, βασίζονται στη διατροφή τους σε προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα χορτονομής όπως επίσης και δημητριακά και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε χημικά για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ζωοτροφών. Εκεί έχει υπάρξει τρομερή πρόοδος τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την κατάσταση όταν γνωρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες της διατροφικές των ζώων και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα της διαδικασίας εκτροφής. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα συνεχίσουμε. Κάποιοι άλλοι ομιλητές έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με την εγκυρότητα των στοιχείων για τις κλιματολογικές αλλαγές. Εγώ, Πρόεδρε, δεν είμαι ειδικό. Δεν είμαι ειδικό στα του κλίματος, εγώ ασχολούμαι με την ε, παραγωγή τη ζωική. Αλλά παρόλα αυτά οι απορίες οι οποίες εξετέθησαν αφορούν ακριβώς το τι εμείς πιστεύουμε γύρω από το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι η απάντηση θα δοθεί μόνο όταν όλοι πάρουν μέρος στη συζήτηση που πρέπει να προηγηθεί και πρέπει να γίνει. Δηλαδή στην παρούσα φάση πρέπει να περιμένουμε τον κόσμο να εφαρμόζει, το κοινό να εφαρμόζει λύσεις μόνο όταν οι λύσεις αυτές είναι χρήσιμες για όλους τους εμπλεκομένους. Μόνο όταν είμαστε σίγουροι για τις τεχνολογίες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι ε, ωφέλιμες για όλους. Θα ωφελήσουν δηλαδή και το σύστημα γεωργικής παραγωγής και τη μείωση της εκπομπής αερίων. Μόνο τέτοιου είδους λύσεις θα μπορέσουμε αν θέλετε να τις ε, ε, πουλήσουμε σε εισαγωγικά και να τις καταστήσουμε αποδεκτές από το ευρύ κοινό. Κάποια μέλη μου ζήτησαν να ιεραρχήσω λίγο τις καλύτερες δυνατές υπάρχουσες λύσεις. Λίγες από αυτές τις λύσεις πράγματι μπορώ να τις ορίσω. Μπορούμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των συστημάτων μας ή να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν έχει σχέση ο τίτλος. Αυτό που σημαίνει είναι το να διαχειριστούμε τα γεωργικά συστήματα παραγωγής με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με το input το οποίο παίρνουν και να μπορέσουμε έτσι να βελτιώσουμε προσωπικά και ποιοτικά το τελικό προϊόν. Σαν παράδειγμα, η σωστή χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων. Είναι συστηματική η προσπάθεια η οποία έχει γίνει για τη μείωση των αζωτούχων στην παραγωγή ε, χορτονομής στην Ιρλανδία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για όλους και για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων, αερίων μάλλον και για τη μείωση του κόστους και για την υγεία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, εδώ έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με καλό τρόπο τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτή θα πρέπει να είναι η κεντρική στρατηγική την οποία οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει βέβαια και τη σωστή διαχείριση των συστημάτων μας. Είτε είναι συστήματα εσοδείας, είτε είναι συστήματα με βοσκοτόπια να βελτιώσουμε την έρευνα και τις επιστημονικές πληροφορίες. Εδώ τίθενται πάρα πολλές επιστημονικού τύπου ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των εδαφών αυτών. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια έχουμε κάνει αρκετά βήματα θετικά σχετικά με την δυνατότητα συγκράτησης και περιορισμού του άνθρακα ε, στις καλλιέργειες ε, είτε σε καλλιέργειες ε, απόδοσης ε, προϊόντων είτε σε καλλιέργειες ε, σε ε, λιβάδια και σε ευοσκοτόπια σε χορτολιβαδικές εκτάσεις εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα πιο συγκεκριμένα θέματα όπως η όπως ε, άλλες λύσεις αφορούν την δυνατότητα χρήσης ψυχανθών σαν παράδειγμα περισσότερος ε, ε, στα, στις χορτολιβαδικές εκτάσεις και νέες τεχνολογίες οι οποίες προς το παρόν δεν είναι βέβαια απόλυτα πρακτικές και εφαρμόσιμες. Η βελτίωση της παραγωγικότητας και η εκτροφή των ζώων είτε μέσα από κανονικές στρατηγικές είτε ε, με συγκεκριμένες στρατηγικές για μείωση ε, ε, αερίων είναι ο βασικός στόχος. Και ένας άλλος τομέας ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η ικανότητα μείωσης των εκπομπών από πλευρά των ζώων μέσω κάποιων παρεμβάσεων, και το λέω αυτό σε εισαγωγικά, που θα τροποποιούν την παραγωγή κρέατος ιδιαίτερα από μυρικαστικά και όταν λέω παρεμβάσεις δεν αναφέρομαι μόνο σε χημικές παρεμβάσεις. Αλλά ίσως να χρησιμοποιήσουμε ε, κάποιες νέες ε, δυνατότητες βιολογίας και γενετικής δυναμικής έτσι ώστε η δυνατότητα χρήσης ας πούμε κάποιων αναστολέων για τη μείωση των υποπροϊόντων της διαδικασίας εκτροφής. Αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό για όλους. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση και της καταναλούμενης ενέργειας γιατί ξέρουμε ότι το μεθάνιο το οποίο παράγεται είναι ενέργεια η οποία χάνεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε μεγαλύτερο κέρδος από την εκτροφή τα όλα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει 10 με 15 χρόνια πριν μπορέσουμε με συστηματικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε. Συγγνώμη αλλά μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα θα ήθελα να απαντήσει ο κύριος Κουκ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία. Αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω στην ομιλία μου είναι να δώσω μία έμφαση στα πολλαπλά ωφέλη που θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε από μία αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τα ευεργετήματα αυτά δεν αφορούν μόνο την άμβληση της κλιματικής μεταβολές αλλά και την βιοπικιλότητα και τα δημόσια αγαθά. Και ένα από τα ερωτήματα είναι ποια είναι τα... τι γίνεται με το γρήγορο κέρδος. Ε από τα γρήγορα φέλη, συγγνώμη. Ένα άμεσο όφελος είναι η μείωση των εκπομπών. Υπάρχει μια εξοικονόμηση του κόστους για τον καλλιεργητή, για τον καλλιεργητή και ε, μείωση της μόλυνσης και ένα όφελος ε, ε, τη μείωση του κόστου καταπολέμησης της ε, επίσης ε, ένα όφελο σε σχέση με τη χρήση των λοιπασμάτων και όπως είπα τη βελτίωση της βιοπικιλότητας. Ένα ερώτημα τέθηκε για τα δημόσια αγαθά και για το κατά πόσο οι καλλιεργητές μιλούν αυτή τη γλώσσα και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν. Η άποψή μου είναι αν θέλουμε να έχουμε μια κοινή πολιτική γεωργίας όπου οι δημόσιες πληρωμές συνδέονται ακριβώς με την παραγωγή δημοσίων αγαθών οι πολιτικοί θα άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτή την γλώσσα, να χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους. Υπάρχει ξεκάθαρα μία ανάγκη μιας μεγαλύτερης μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων προς αυτούς που διαχειρίζονται τη γη. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο έχει θέσει κλειδί εδώ. Επίσης ασχοληθήκαμε με το θέμα των εκπομπών του άνθρακα και τις ε, παραγωγής του άνθρακα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Νομίζω ότι εδώ δεν θα πρέπει να εξαγάγουμε τα δικά μας προβλήματα προς τα έξω. Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τη δική μας γεωργία με ένα βιώσιμο τρόπο, ούτως ώστε να διαφυλάσσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση για το τι είδους γεωργία θα έπρεπε να έχουμε και πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ερώτημα εδώ δεν υπάρχει μία μοναδική ερώτηση αλλά νομίζω το είδους γεωργίας που θα έπρεπε να έχουμε είναι αυτό που συνάδει με τη φύση ε, που θα υποστηρίζει το έδαφος δηλαδή να μην ε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη φύση του εδάφους ή τη φύση του κλίματος, να αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους δηλαδή. Κανείς από εμά σήμερα δεν αναφέρθηκε στο ακόλουθο ε, θέμα και δεν ξέρω αν θα αναφερθεί στις επόμενες παρουσιάσεις. Πρόκειται για τη σημασία του ύδατος στις, ε, στην κλιματολογική αλλαγή. Νομίζω ένα θέμα στο οποίο δεν δώσαμε αρκετή προσοχή. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνώμονές μας και συνεχίζουμε την ακρόαση με τις επόμενες παρουσιάσεις τους οποίους ε, ευχαριστούμε προκαταβολικά για την παρουσία του σήμερα εδώ. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Σαντόφσκι που θα μιλήσει για σενάρια της αλλαγής του κλίματος για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και πολιτικές επιλογές στο πλαίσιο της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Ο κύριος Σαντόφσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκδήλωση αυτή. Δεν ε, σας κρύβω ότι Υπάρχει βεβαίως κάποια ε, επιφύλαξη στις αντιδράσεις και στα, στα όσα ακούμε και στα επιχειρήματα που προβάλλονται γιατί πολλές φορές προετοιμαζόμαστε για πράγματα που μπορεί να μην συμβούν. Σημαντικό πάντως είναι να έχουμε ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τις κλιματικές μεταβολές και διακυμάνσεις μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα μιλάμε για την ε, μείωση, άμβλυνση των ε, κλιματικών επιπτώσεων. Ακούσαμε λεπτομερείς πληροφορίες ε, επί του θέματος αυτού σήμερα. Ας δούμε τον καιρό στην Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία μπορούμε να επιστήσουμε την προσοχή. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε τη βροχόπτωση στο τέλος του αιώνα και υπάρχουν και κάποια άλλα ε, στοιχεία που περιλαμβάνονται και μπορεί να αλλάξουν ανάλογα αν εξετάζομαι το βόρειο ή το νότιο τμήμα της Υπήρου. Τώρα, το πρόβλημα που συζητούμε σήμερα είναι οι εκπομπές και προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε το ποσοστό που προέρχεται από τη γεωργία. Είδαμε ότι οι συνολικές εκπομπές από τη γεωργία είναι περίπου το 9%. Τώρα, το επόμενο ερώτημα πρέπει να είναι αν όντως η γεωργία ε, είναι υπόλογη για αυτό το ποσοστό των αλλαγών, γιατί είναι δύσκολο να ξέρουμε ποιο κομμάτι από αυτό είναι ανθρωπογενές, ποιο είναι, προέρχεται από, και οφείλεται ε, στη, ε, στη φύση. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε προσεκτικά στις ε, ε, εξετάσεις μας για να μην κάνουμε μεγάλα λάθη. Για παράδειγμα, αν δούμε την εντερική ζύμωση και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων, αυτό είναι τμήμα του κύκλου της ενέργειας στη γεωργία. Δείτε εδώ κάποια στοιχεία με τα αέρια θερμοκηπίου. Η γεωργία πάλι αναφέρεται με το 9% στη συνολική πίτα. Είναι σημαντικό όμως να δούμε σχετικά τα νούμερα αυτά ε, και σε σχέση με τις εκπομπές από άλλες πηγές. Πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε με μια προοπτική αυτά και να ε, ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που δεν θα οδηγήσει ε, σε πράγματα για τα οποία θα μετανιώσουμε. Ε, μπορεί να οργανώσουμε τις προσεγγίσεις μας έτσι ώστε να ωφεληθεί η Γεωργία. Η εταιρεία McKenzie διεξήγαγαν μια έρευνα στην Πολωνία με σκόπο τη μείωση των εκπομπών. Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς όπου είναι δυνατόν να έχουμε μείωση με συγκεκριμένο κόστος. Είναι σημαντικό να το δούμε και το κόστος, αλλά υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Τώρα, αν θέλουμε να εξετάσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, εδώ θα πρέπει να δούμε την λειψιδρία, τις ξηρασίες. Έχουμε δει ε, τέτοια προβλήματα. Είναι σημαντικό να δούμε ολόκληρη, συνολικότερα, την οικονομία του ύδατος. Επίσης ε, υπάρχουν επιδράσεις ε, με την έννοια νέων φυτικών νόσων, ε, ζυζάνια, για παράδειγμα που πλήττουν την πατάτα. Αυτό συνέβη στην Πολωνία. Αναφέρεται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση στην παραγωγή της πατάτας κατά 40% στην Πολωνία ακριβώς λόγω των ε, προβλημάτων αν τα αφήσουμε να συνεχιστούν. Έχουμε ε, μείωση της παραγωγής λοιπόν, ε, προβλήματα λόγω της αύξησης θερμοκρασίας στα ζώα, αυξημένο στρες και πολλές φορές πρέπει να λάβουμε υπόψη στα κρέα καιρικά φαινόμενα ή την ε, καταλληλότητα των καλλιεργειών που πρέπει να ε, είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Πολλές φορές η αύξηση της θερμοκρασίας ε, είναι αποτρεπτική για ορισμένες καλλιέργειες, όπως και η λειψιδρία που περιορίζει την παραγωγή σε πρώην σχεδόν αποκλειστικά αγροτικές περιοχές. Μπορούμε να κάνουμε προβολές ε, μέχρι το 2080 και κάνοντας συγκρίσεις με την περίοδο 61-90. θα συνεχιστούν από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα λειψιδρίας, προβλήματα άρδευσης και πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό η αγροτεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε λύσεις εδώ. Εδώ είναι ο χάρτης καλλιεργειών της Ευρώπης και αν δείτε την απόδοση από τις καλλιέργειες βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές ε, και στο βορρά και στο νότο της Ένωσης. Ποια είναι για μας τα κέρια προβλήματα. Οι πολιτικοί και οι γεωργοί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές όπως αυτές που αναφέρονται μπορεί να λάβουν χώρα και είναι σημαντικό να είναι προετοιμασμένοι. Οι γεωργοί βέβαια είναι εκείνοι που θα πληγούν, θα επηρεαστούν και οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν τη ζωή τους την ίδια. Βέβαια οι γεωργοί ε, συμφωνούν με τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, άλλωστε δεν μπορούν αλλιώ να επιβιώσουν. Βέβαια η προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνολογίες και η υποδομή. Η... Ο γεωργικός πληθυσμός πάντως πρέπει να είναι ενήμερος, να γνωρίζει να έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη και τον τρόπο για τις αλλαγές. Χρειάζονται υποστήριξη λοιπόν οι γεωργοί για να ξέρουν πώς θα προσαρμόζονται. Είναι ευπροσάρμοστοι και το έχουν αποδείξει, αλλά θα πρέπει να καθοδηγηθούν ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν με βάση τις διαθεσιμότητες. Είδατε το χάρτη της Ευρώπης πολλές φορές, όμως οι απαντήσεις είναι τοπικές, περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών. Οι ε, μονοσήμαντες προσεγγίσεις ε, είναι επιζήμιες. Θα πρέπει να δούμε και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε υποεθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν εδώ κάποιες ε, παύλες ε, που αφορούν τις συστάσεις για τη μείωση των αρνητικών ε, φαινομένων. Είναι σημαντικό αυτό και για την δυνατότητα προσαρμογής. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μακροπρόθεσμη πολιτική μπορούμε να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020 και να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την ευελιξία των γεωργών, ε, ιδιαίτερα ε, όταν πρόκειται για την ε, διαχείριση των υδάτων. Θα πρέπει η διαχείριση των εκμεταλλεύσεων να προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και κάτι άλλο πρέπει να προσθεθεί εδώ που αναφέρθηκε στη συζήτηση και που θα παίξει κύριο ρόλο στο μέλλον. Αν θέλουμε να έχουμε ε, γεωργία στο σωστό επίπεδο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει έλλειψη γης. Και κάποια στιγμή υπάρχει σύγκρουση μεταξύ γεωργίας από την άλλη και περιφερειακής πολιτικής Πρέπει λοιπόν στο μέλλον να εξευρεθούν περισσότερες υγιές για να διατηρηθούν τα επίπεδα παραγωγής ε, που έχουμε συνηθίσει ε, να έχουμε. Εδώ οι επιστήμονες μπορούν να βοηθήσουν αναπτύσσοντας νέες καλλιέργειες, είδη και ποικιλίε. Νομίζω ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις ε, από όλα αυτά και για την κοινή αγροτική πολιτική. Η ΚΑΠ δεν μπορεί ε, πρέπει βράχει πρόθεσμα να προβεί στη λήψη μέτρων για την ε, μείωση πολλών ε, αρνητικών φαινομένων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα του κλίματος στη Γεωργία. Ε, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας ορθές πρακτικές που μειώνουν τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής με τη χρήση νέων μέσων, ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει μια σχέση μεταξύ ε, του, του, του, της επιστημονικής κοινότητας και των γεωργών της ε, άσκησης της γεωργικής πολιτικής επίσης. Πρέπει να υπάρχει ε, αλληλεπίδραση. Ε, η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ καλό παράδειγμα για την ενημέρωση διαφορετικών τομέων της κοινωνίας μας. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη γιατί οι περισσότεροι σκέφτονται καλύτερα από τον ναι, έναν. Ευχαριστώ. και εγώ τον κύριο Σαντόφσκι. Ο πέμπτος εμπειρογνώμων που θα ακούσουμε σήμερα είναι ο κύριος Γιάν Φερχάγκεν. Είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Βάχενιγχεν στην Ολλανδία. Θα μας μιλήσει για την προσαρμογή της γεωργίας στις κλιματολογικές αλλαγές και τι συνέπειες θα έχει κάτι τέτοιο στην ΚΑΠ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω προετοιμάσει την παρουσίασή μου στα αγγλικά, αλλά είδα ότι μπορώ να μιλήσω την Ολλανδική και συνεπώς θα συνεχίσω σε αυτή. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις δυνατότητες προσαρμογής της γεωργίας στις κλιματολογικές αλλαγές και θα προσπαθήσω να το συνδέσω με την ΚΑΠ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι οι κλιματολογικές αλλαγές είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με συνέπειες οι οποίες κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν άλλες περιοχές του κόσμου οι οποίες φύγονται από τις κλιματολογικές αλλαγές πολύ χειρότερα από ό,τι η Ευρώπη. Η Ποσαχαρική Αφρική σαν παράδειγμα στην, στην ε, Ευρώπη συγγνώμη, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο βόρειο τμήμα και το νότιο τμήμα ε, πόσο μάλλον σε περιοχές του κόσμου όπως η Αυστραλία όπου τα θέματα είναι πάρα πολύ ε, σοβαρά. Υπάρχουν σε περιοχές του κόσμου ήδη άμεσες συνέπειες στην παραγωγή, στην παραγωγή φυτών, ε, φυτικών προϊόντων ή ζωικών προϊόντων. Μείωση της βροχόπτωσης, υψηλότερες θερμοκρασίες. Απ' την άλλη υπάρχουν και κάποιες ε, λιγότερο γνωστές ε, θετικές συνέπειες σε ορισμένες περιοχές σαν παράδειγμα έχει επιβληθεί αν θέλετε η καλύτερη διαχείριση των ε, υδάτινων πόρων. Και νομίζω ότι έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο ε, τις συνέπειες των ακραίων φυσικών φαινομένων όπως το χαλάζι, οι καταιγίδε, η ξηρασία. Γενικά έχουμε αποκτήσει μια τεχνογνωσία ε, για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Υπάρχουν πάντως προβλήματα όπως ε, η αύξηση του επίπεδου της θάλασσας, η σχόρηση ε, του θαλασσινού νερού στους υδάτινους πόρους και ο κίνδυνος επίσης ασθενειών και επιδημιών που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω ακριβώς της αύξησης της θερμοκρασίας. Ο άνθρωπος φυσικά παίζει τον κυρίαρχο ρόλο αλλά παρόλα αυτά οι επιπτώσεις αυτές αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του πλανήτη. Επηρεάζονται φυσικά και οι τιμές των προϊόντων εφόσον τα προβλήματα αυτά μονιμοποιούνται. Υπάρχουν επίσης βλάβες οι οποίες προκαλούνται από τα φυσικά φαινόμενα στις υποδομές, στα κτίρια, ε, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε ορισμένες περιοχές του κόσμου από τις συστηματικές πλημμύρες, από τις χαλαζοπτώσεις Συνεπώς η γεωργία και οι κλιματολογικές συνθήκες συνδέονται άμεσα γιατί η γεωργία υπόκειται φυσικά σε καθημερινή φάση στον έλεγχο του κλίματος. Εφόσον λοιπόν η γεωργία πρέπει και μπορεί να προσαρμοστεί, αυτό θα έχει άμεσες συνέπειες γενικότερα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μετριασμό συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών μια ε, σταθερή και, κλιμα... και φιλική προς τις αλλαγές του περιβάλλοντος πολιτική νομίζω ότι ε, θα ωφελήσει τους πάντες. Υπάρχουν ε, βέβαια συνέπειες και σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίσης επίπεδο Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, να εντάξουμε τις κλιματολογικές αλλαγές στα γεωργικά προγράμματα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί μια υψηλή δόση προσαρμοστικότητας. Με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζονται οι συνέπειες αυτές ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με την περίπτωση τι αλλαγές ε, καλείται να επιφέρει στον τρόπο παραγωγής ο καλλιεργητής. Αυτό συνδυάζεται και με άλλα προβλήματα όπως η έλλειψη διαδοχής στις γεωργικές καλλιέργειες στη Βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ολλανδία. οι κλιματολογικές και οι οικονομικές συνθήκες είναι απαραίτητες για να ληφθούν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα, είτε σε επίπεδο επιχειρηματικότητα στην Γεωργία, είτε σε επίπεδο λήψης πολιτικού τύπου αποφάσεων. Κάναμε κάποιες μελέτες λοιπόν για τις συνέπειες των αλλαγών αυτών στις γεωργικές αγορές, ιδιαίτερα για τις βόρειες επαρχίες των κάτω χωρών, να εξετάσαμε τις αλλαγές στον τομέα της παραγωγής, στον τομέα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είδαμε το ποια είναι η ζήτηση, σε τι επίπεδο παραμένει η ζήτηση, αν απαιτείται περαιτέρω αύξηση της παραγωγής και έχουμε καταλήξει σε δύο σενάρια, στο α και το β. Το α είναι το σενάριο που καλύπτει αυτά τα οποία χρειάζεται η ανοιχτή αγορά και το δεύτερο σενάριο είναι αυτό το οποίο θα ονόμαζα το σενάριο του περιφερειακού προστατευτισμού. Είναι λίγο δυσνόητα ίσως όλα αυτά, αλλά και στην Γαλλία όπως βλέπουμε εδώ και στη Σουηδία έχουν γίνει αντίστοιχες μελέτες. Στο κάτω μέρος βλέπετε στην αριστερή πλευρά μηδενικές συνέπειες για το σύνολο της Ευρώπης. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη μας την αύξηση εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, υπάρχουν μερικές φορές και θετικά αποτελέσματα που οδηγούν στην αύξηση των βροχοπτώσεων. σε επίπεδο τεχνολογιών τις οποίες χρησιμοποιούμε. Βλέπετε τα τέσσερα σενάρια τα οποία είναι διαθέσιμα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δύο πρώτα. Λέει. Οι κλιματολογικές συνέπειες έχουν άμεσες συνέπειες στην απόδοση της ε, εσοδείας Γίνονται οι έρευνες, συνεχίζονται οι έρευνες οι οποίες θα μας οδηγήσουν ελπίζουμε σε περισσότερες γνώσεις σχετικά με την αύξηση της παραγωγικότητας. Το δεύτερο σενάριο δείχνει ότι οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πλέον, είναι πλέον δεδομένες αλλά είναι αυτό που θα έλεγα πιο αργές, ιδιαίτερα στα δημητριακά. Στα δημητριακά και σχετικά με την παραγωγικότητα γύρω από τα δημητριακά. Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τη δεκαετία του 1990 μπορούμε να ξέρουμε ε, το τι θα συμβεί στο μέλλον σε ένα προβλεπτό μέλλον, όχι βέβαια στο 2050. Φαίνεται να υπάρχουν βελτιώσεις πάντως σε ορισμένες τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες μέσω της χρήσης και διαφορετικών τεχνολογιών. Αν δει κανεί ε, τη ζήτηση και την προσφορά για τα δημητριακά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δει κανεί ότι θα υπάρξουν λιγότερες εισαγωγές γιατί δημιουργούνται δυνατότητες μεγαλύτερης εσωτερικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα οφείλεται γιατί θα υπάρξει αύξηση των βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές. Αυτά στο σενάριο Α1. Στο σενάριο Β2 βλέπει κανείς ποιο είναι το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται. Μια αύξηση της παραγωγής μπορεί να λειτουργήσει ρυθμιστικά για μια μακροπρόθεσμη μεγαλύτερη χρονική περίοδο σε σχέση με το ε, μοντέλο Α1, το σενάριο Α1. Πάντως υπάρχουν διακυμάνσεις ε, σε σχέση με την παραγωγή ανάλογα με τις περιοχές. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η πυκνότητα του πληθυσμού και διαφορετικά στοιχεία φυσικά παίρνουμε για περιοχές οι οποίες είναι γεωργικές, χαρακτηρίζονται σαν γεωργικές περιοχές και άλλες μη γεωργικές ή περισσότερο αστικές. Βλέπετε ότι για το σενάριο Α1 για το 2050 μέχρι το 2050 θα υπάρχει αύξηση παραγωγής τσίτου δημητριακών ιδιαίτερα στην βορειοδυτική Γαλλία η οποία είναι η μεγάλη θα έλεγα σιτοπαραγωγός ευρωπαϊκή περιοχή η Μπος. Και αυτό θα έχει θετικές συνέπειες και για άλλες περιοχές της Ευρώπης. Θα υπάρξουν αλλαγές και στο εσωτερικό των διαφόρων χωρών βλέπετε ότι υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις οι οποίες ε, μάλιστα είναι μεθοριακές ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες χώρες και εκεί ακριβώς απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και προγραμματισμός. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τελικά είναι σημαντική η κλιματολογική αλλαγή για τις ε, δυνατότητες προσαρμογής και μετριασμού στην γεωργίας Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί για να μην πω και περισσότερο σημαντικοί. Εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση ε, το πόσο θα επηρεαστεί από τις κλιματολογικές αλλαγές. Η τεχνολογική πρόοδος απαιτεί να υπάρξει έρευνα και ανάπτυξη περισσότερη από ό,τι σήμερα και χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογή για να δούμε τι συνέπειες θα υπάρξουν για τις ε, ε, πολιτικές μετρίεσης των αρνητικών συνεπειών. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές, τι μπορούμε να συγκρίνουμε, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τις εμπειρίες άλλων θα υπάρξουν αλλαγές σε ορισμένες περιοχές ακόμα και για την αλλαγή του εξοπλισμού, του μηχανολογικού ο οποίος χρησιμοποιείται, ελκυστήρες, οχήματα κτλ. θα πρέπει να δούμε και τρόπους ακόμα καλύτερης ανταπόκρισης και αντιμετώπισης των συνεπειών ακραίων φυσικών φαινομένων. Θα πρέπει να δούμε το κόστος συνολικά της αντιμετώπισης των συνεπειών δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς το κόστος αυτό των μέτρων προσαρμογής και μετρίασης των συνεπειών παραμένει ένα ανοιχτό θέμα. Υπάρχουν φυσικά και ειδικέ συνέπειες περιφερειακού χαρακτήρα στο εσωτερικό, οι οποίε μπορούν να ληφθούν υπόψη στο εσωτερικό της κοινή αγροτικής πολιτικής. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει νομίζω συνολικά τον προγραμματισμό της ΚΑΠ και θα καταστήσει ε, πιο ε, συμβατές με το περιβάλλον της διαδικασίας παραγωγής. Als je alles lokaal En toch, de laatste weer. Ja, ik ben onderzoeker. Ik vind het toch wel leuk om dat iedere keer te noemen. Het is toch en blijft een belangrijke. Want er zit een kostenplaatje aan, ook in het voortraject. En dat zijn investeringen die toch redelijk lang kunnen... Αυτό το οποίο έχει σημασία τελικά είναι το τι επενδύσεις μπορούμε να προβλέψουμε μακροπρόθεσμα για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών συνεπειών. Οι νέες τεχνολογίες διαρωτώμεθα μπορούν να, προσ... να λειτουργήσουν σαν παράγον επιτάχυνσης των αλλαγών. Υπάρχει δυνατότητα να επιταχύνουμε τις προθεσμίες. Σε δέκα χρόνια χρειάζονται για να καλλιεργηθεί μια νέα ποικιλία του σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάγκεν. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρώτα έχει το λόγο η κυρία Πάλσεν. Ήταν, ε, άκουσα με μεγάλη μου χαρά τους εμπειρογνώμονε σήμερα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεφόλ για την εξαιρετική του έκθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο της εικόνας. Πριν ξεκινήσουμε με τη συζήτηση των επιμέρους πτυχών, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε σύμφωνα με αυτές τις βασικές γραμμές ε, σκέψης όταν ασχολούμεθα με τις λεπτομέρειες, όταν περάσουμε στις λεπτομέρειες που στον ουρανό, για να πούμε πού στον ουρανό τοποθείται το αστέρι που κοιτάζω αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να έχουμε το σύνολο του ουράνου θόλου για να εντοπίσουμε τις λεπτομέρειες. Η δασοκομεία και η γεωργία δεν είναι πρόβλημα στις κλιματολογικές αλλαγές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο θέμα των εκπομπών αερίων, αλλά θα πρέπει μάλλον να εξετάσουμε την ικανότητα του εδάφους και των δασών να παγιδεύουν, να δεσμεύουν τον άνθρακα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ και αν ε, εξετάσουμε πράγματα από αυτή την οπτική γωνία θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα. Όχι μόνο η παγίδευση του άνθρακα, αλλά μπορούμε να πάμε πολύ μακρύτερα. Εάν διαχειριστούμε τη γεωργία με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα θα έχουμε βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, θα έχουμε καθαρότερη ατμόσφαιρα, θα έχουμε μια βελτίωση της βιοπικιλότητας, θα είμαστε σε θέση να επιλύσουμε μία σειρά θεμάτων προσπαθώντας να εξεύρουμε μεθόδους γεωργικής παραγωγής που εξετάζουν το έδαφος, φροντίζουν το έδαφος μάλλον και νομίζω ότι θα σεβαστούμε τον τρόπο που θα προστατεύσουμε τη μητέρα γη. Είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την, ε, το παραγωγικό μας δυναμικό. η αεροτρέα, ε, τα αεροτρέα εδάφη θα αποφέρουν καλύτερη σοδιά εάν έχουν βελτιωμένο φυσικό περιβάλλον, ένα υπέδαφος ε, βιώσιμο. Εάν δεν εξετάσουμε λοιπόν τη συνολική εικόνα θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι δεν θα πιστεύουν στη διασύνδεση μεταξύ εκπομπών αρίων θερμοκηπίου και κλιματολογικών αλλαγών. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι ατυχέ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η μεταβολή του κλίματος είναι ένα γεγονός Και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στις μελλοντικέ μας σκέψεις για την γεωργία, για την γεωργική πολιτική. Μία λεπτομέρεια που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική αλλαγή είναι η εξής. Εάν χρησιμοποιήσουμε τις ε, παρούσες τεχνικές για τη δασοκομεία και τη γεωργία, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την, ε, με τον τρόπο αυτό την ε, αυτό, συντηρούμενη ενέργεια. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας λοιπάσματα και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλοιπα της ε, σοδιάς ε, χρησιμοποιώντας βιοαέριο και λοιπά ενεργειακά κύτταρα. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και τα ε, άλλα είδη καταλήπων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε, όπως σας είπα, την συνολική εικόνα και να, στη συνέχεια να εντοπίσουμε τις λεπτομέρειες. Τι είδου ε, ε, γεωργία επιθυμούμε, θα είναι εντατική, βιολογική κλπ. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι καμία από τις ε, παρούσες μεθόδους είναι απολύτως εφικτή για το μέλλον από μόνη της. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε μάλλον είναι ένας έξυπνος συνδυασμό των παλαιών και νέων μεθόδων. Υψηλή τεχνολογία, και ε, βιολογικές, σε συνδυασμό όμως με τις ε, βιολο, λεγόμενες βιολογικές ε, μεθόδους, τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας. Δεν νομίζω ότι κανείς μέχρι στιγμής έχει εξετάσει σοβαρά αυτή τη δυνατότητα. Αλλά και πάλι σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ο Ζωζέ Μποβέ έχει το λόγο. Ναι, θα ήθελα να επανέλθω στις προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σήμερα γιατί πιστεύω ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό στην έκθεση και αυτό, το αυτό που υπογραμμίζει ο Στεφάν Λεφόλ είναι όταν λέει ότι η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να είναι αποδοτική από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για το ένα θέμα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και τα άλλα θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό το οικονομικό όραμα και νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να καταδείξουμε ότι οι λύσεις δεν είναι ασύμβατες μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Δεν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν συστήματα σήμερα τα οποία είναι επιβλαβή από οικολογική άποψη και από οικονομική άποψη δεν είναι κατά ανάγκη αποδοτικά. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το υπερβολικό βιομηχανικό μοντέλο πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Στη Γαλλία έχει γίνει μια έρευνα και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ότι έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Γεωργίας για την δυνατότητα αναπροσανατολισμού ενός τμήματος των γεών ε, σε καλλιέργειες ψυχανθών. Στη Γαλλία σήμερα ε, υπάρχουν ε, ε, υπήρχαν το 1963 εκατομμύρια γες με καλλιέργειες ψυχανθών. Σήμερα υπάρχει μια σημαντική μείωση. Ταυτόχρονα υπάρχουν εισαγωγές σόγιας και βρισκόμαστε σε μια ισορροπία που είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή από τη μία μπορούμε να μειώσουμε το 41% αυτών των εισαγών με μια κανονική αύξηση της τάξης του 7% των ψυχανθών στις καλλιέργειες με σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων και την παγίδευση του διοξιδίου του άνθρακα. Και ε, μπορούμε να φτάσουμε οικονομικά να πετύχουμε. Αυτό το οποίο χάσουμε από τις εισαγωγές των δημητριακών θα το κερδίσουμε από την μείωση του κόστους των λιπασμάτων και από τα κέρδη της αποθήκευσης του άνθρακα σήμερα το να λέμε ότι θα κάνουμε μια γεωργία που είναι συμβατή με το περιβάλλον δεν σημαίνει ότι είναι μια γεωργική πολιτική αντιοικονομική. Αυτό είναι ο ισολογισμό που θα ήθελα πραγματικά να υπογραμμίσω για να πάμε στην κατεύθυνση της προσαρμογής ε, από τη μία, αλλά ταυτόχρονα το θέμα των σπόρων που είναι μια διαδικασία η οποία ε, έχει ένα μέλλον. Ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης των σπόρων μελλον ο καλυτερο τροπο βελτιωση των σπορων ειναι να συμμετάσχουν ήδη οι καλλιεργητές στις έρευνες, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να προσφέρουν εδώ τις καλύτερες ιδέες όσον αφορά την αλλαγή των ε, σπόρων, τη βελτίωση των σπόρων. Ευχαριστώ κύριε Σεκέρσκι. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις, ή σχόλια μάλλον, αν μου επιτρέπετε ακούγοντας σήμερα τους ε, εμπειρογνώμονες, ακούγοντας και τον εισηγητή, ερωτώ ποια είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Από πού θα έχουμε την καλύτερη απόδοση των επενδύσεών μας. Μιλάμε για προσαρμογή, ενέργεια, έρευνα, γεωργία Όλοι αυτοί είναι τομείς. Ε, πού πρέπει να κάνουμε λοιπόν την ε, οικονομική μας αυτή προσπάθεια, πού πρέπει να επενδύσουμε. Είναι σημαντικό αυτό και για το Κοινοβούλιο. Ε, τώρα, για την εντατική παραγωγή. Έχουμε πείρα πολλών ετών. Ξέρουμε δηλαδή ε, τα υπέρ και τα κατά εκτατικής και εντατικής καλλιέργειας. Η ισορροπία των δύο θα επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. Είναι δυνατόν να ε, δούμε ποια κλίμακα παραγωγής θα αποβεί προσοδοφόρα λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της βιολογικής γεωργίας μεταξύ άλλων. Πρέπει να εξετάσουμε διάφορα είδη γεωργίας, νομίζω, ε, ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, για να αποφασίσουμε αν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και την οικονομία του ύδατος. Μέσα σε 10 χρόνια είδαμε μεγάλη αύξηση της ε, γεωργίας, της βιολογικής γεωργίας. Αυτό είναι σαφής τάση, την είδαμε. Τώρα θα πρέπει να καταδείξουμε πόσο σημαντική είναι η ΚΑΠ ως πολιτική, πόσο σημαντική είναι για την κοινωνία, τους καταναλωτές, το περιβάλλον. Πρέπει να δούμε και την περιβαλλοντική διάσταση. Καμιά φορά παραμελούμε παραγνωρίζουμε το ζήτημα της ασφάλειας στην παροχή τροφίμων. Καμιά φορά ξεχνάμε ότι η ΚΑΠ ε, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε και μας τροφοδοτούσε με τρόφιμα. Το 2007 και μετά ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε, στον τομέα του κόστους των τροφίμων και της παροχής τροφίμων. Και βέβαια ε, η Γεωργία ξαναβγήκε στο προσκήνιο και στα πρωτοσέλιδα μετά από κάποια χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο γρήγορες ερωτήσεις μια γραφική παράσταση στην αρχή ήταν πολύ τρομακτική γιατί έδειχνε πρόβλεψη βροχοπτώσεων τα επόμενα 70 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο που μας τα έδειξε αυτά πόσο βέβαιος είναι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο γιατί δεν είναι καθόλου αξιόπιστες οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις γιατί αν γίνει αυτό θα υπάρξουν κύματα μεγάλα μεταναστευτικά ε, προς τα υγρά κλίμακα ή από τα υγρά κλίματα. Θα συμβεί αυτό. Κάποιος άλλος ομιλητής μίλησε για την πατατοπαραγωγή σήμερα στην Πολωνία. Οι τελευταίες τάσεις ε, δείχνουν ότι έχει γίνει ψυχρότερο το κλίμα. Αυτό εννοεί που, και όταν λέει ότι θα επηρεαστεί η παραγωγή της πατάτας στην Πολωνία. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Ίσως η έμφαση στην κλιματική αλλαγή μας αποπροσανατολίζει από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων Χρειαζόμαστε ως κοινοβούλιο, χρειάζεται ως κοινοβούλιο να δούμε το θέμα αυτό, γιατί συμφωνούν οι επιφυλακτικοί για την κλιματική αλλαγή, αλλά και αυτοί που την πιστεύουν, όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Οπότε έχουμε έναν κοινό που παρονομαστεί. Μην πολωνόμαστε, ας δούμε που, εκεί όπου συμφωνούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, δεύτερον, μία παρατήρηση που ανέφερε ο τρίτος ομιλητής για τα προγράμματα που το πρόβλημά τους είναι ότι καμιά φορά έχουν ασυνέχεια. Καμιά φορά τα ωφέλη των προγραμμάτων σταματούν μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και αυτό θα πρέπει να το δουν οι ειδικοί. Συγκεκριμένο ερώτημα για την άρρωση των εδαφών. Γιατί υπάρχει αντίσταση στην ελάχιστη καλλιέργεια. Η εμπειρία μας στην Ιρλανδία ήταν μεικτή αλλά δεν ε, σπέβδει κανείς προς αυτή την κατεύθυνση. Οι γεωργοί δεν είναι ανόητοι. Θα πρέπει να τους πείσουμε ε, όταν ε, για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι δεν αξιοποιούμε την καλύτερη γνώση που έχουμε. Δεν την εφαρμόζουμε στις εκμεταλλεύσεις. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη γεωργία σε πολλά κράτη-μέλη τώρα ε, εξαντλούν το έργο τους συμπληρώνοντας έντυπα για τους αγρότες χωρίς να δίνουν συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση των εδαφών. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε επίπεδο πολιτικό τέλος κανείς δεν μίλησε για την κερδοφορία της γεωργίας, γιατί αν δεν βγάζουν κάποια εισόδημα οι αγρότες δεν θα ενδιαφερθούν για τίποτα ούτε θα έχουν τα λεφτά για να επενδύσουν στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών κλπ. κλπ. Θα ήθελα τα σχόλιά σας επί αυτών. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Χάουσλινγκ. Παρακαλώ. Ναι. Ε, ναι. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, προηγούμενες ε, συζητήσεις. Αυτό το οποίο με κατέπληξε ήταν ότι από ορισμένους τίθεν αφιβόλω ορισμένα δεδομένα. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάποιες ε, παρατηρήσεις ως γνώμονα των αναλύσεων μας, αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Δηλαδή ε, υπάρχει μια παγκόσμια τάση η οποία είναι αδιαμφισβήτητη και δεν το έκανε και κανείς από τους επιστήμονες. Και θα πρέπει να αντιδράσουμε ταχαίως σε αυτή την τάση μέσω αναθεώρησης της ΚΑΠ. Η Γεωργία θα πρέπει να προσαρμοστεί φυσικά εδώ. Υπάρχουν στόχοι μείωση που θα πρέπει να εκπληρώσουμε. Και εδώ έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα. Εγώ θεωρώ ενδιαφέρον ότι δόθηκε έμφαση στο γεγονό ότι χρειάζεται να κάνουμε μια βιώσιμη γεωργία, η οποία να είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον, ε, διατήρηση των πράσινων ε, ζωνών σε πολλές χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ε, θα πρέπει να ε, αμφισβητήσουμε την εντατική καλλιέργεια σχέση με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Δηλαδή θα πρέπει ε, επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα ότι μελλοντικά θα, έχουμε, θα πρέπει να υπάρχει μια μείωση των, του των καυσίμων. Δεν είναι να γεωργική πολιτική χωρίς την πτυχή προστασία του περιβάλλοντος. Ε, γι' αυτό θα πρέπει μελλοντικά να φωτίσουμε περισσότερο τις ε, προσεγγίσει που εφαρμόστηκαν σε διάφορε χώρε και στον δεύτερο πυλώνα. Νομίζω ότι σήμερα δεν έγινε αυτό επαρκώς. Θα πρέπει να κάνουμε έναν ε, απολογισμό ε, μέχρι που έφτασαν αυτές οι χώρες, αυτά τα μοντέλα ε, και που θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην γεωργική μας πολιτική. Στα θέματα αυτά θα πρέπει να εμβαθύνουμε μελλοντικά. Συνολικά νομίζω ότι αυτή ήταν μια συζήτηση η οποία θα συνεχίσει να μας συνοδεύει και ελπίζω ο εισηγητής να μπορέσει να συμπεριλάβει πολλά από αυτά τα ερεθίσματα στην έκθεσή του και όπως σας είπα η συζήτηση αυτή θα μας συνοδεύει ασφαλώς και τα επόμενα χρόνια ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις που μας θέσατε. οι συγκητές που μίλησαν στο πρώτο τμήμα της συζήτησης μπορούν να μιλήσουν και τώρα εφόσον το επιθυμούν. Ο κύριος Σαντόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα Ευχαριστώ πράγματι. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ε, απευθύνθηκαν περισσότερο σε μένα. Καταρχάς να πω ότι οι κλιματολογικές αλλαγές είναι ε, ένα ουσιαστικό ε, δεδομένο τώρα πλέον και είναι κάτι το οποίο ε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε παρά κάποιες αμφιβολίες. Βλέπουμε σαν παράδειγμα κάποιες ασθένειες ε, οι οποίες ε, να αυξάνεται η συχνότητά τους, να διευρύνεται η ζώνη στην οποία σημειώνονται οι ασθένειες αυτές, οι ζωονόσοι αυτές και εκεί έχει παίξει ρόλο και η κλιματολογική αλλαγή. Τίθεται επίσης ένα θέμα γενικότερο σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την προστασία του εδάφους. Δεν υπάρχει ουσιαστική τέτοια πολιτική. Υπάρχει συστηματική υποβάθμιση του εδάφους και του επιφανειακού αλλά μερικές φορές και σε μεγαλύτερο βάθος και απώλεια επιπέδων γον, ε, παραγωγικότητας το έδαφος πάβει να είναι τόσο έφορο όσο στο παρελθόν. Απαιτείται λοιπόν μια οικονομική βοήθεια και μια συγκεκριμένη πολιτική. Ένας άλλος τομέας ο οποίος πρέπει να μας απασχολήσει με πολύ πιο έντονο τρόπο είναι οι μεταφορές. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς ε, τις μεταφορές γιατί ο τομέας αυτός είναι τεράστιος και από το μέγεθός του είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπιεστεί. Εδώ τώρα αν εξετάσει κανείς την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας χρειάστηκε να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή θα δει ότι οι συνέπειες δεν ήταν αντίστοιχες όπως επίσης και οι επενδύσεις δεν ήταν αντίστοιχες. Οι πόροι τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας δεν έχουν νομίζω φτάσει στο επίπεδο που χρειάζεται έτσι ώστε να λυθούν προβλήματα τα οποία συνδέονται με θέματα όπως η άρδευση κτλ. σχετικά τώρα με τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών. Κάποιοι ερώτησαν είναι πραγματικές οι επιπτώσεις αυτές. Δεν μιλάμε για προβλέψεις, μιλάμε για σενάριοι. Τι εννοούμε εδώ. Εννοούμε κλιματολογικές αλλαγές οι οποίες είναι δεδομένες, τις διαπιστώνουμε. Δεν κάνουμε προγνώσεις, τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας τις συνέπειες προσπαθούμε να εκτιμήσουμε. Διαμορφώνουμε διάφορα σενάρια όπως είπα και βλέπουμε τι επιπτώσεις υπάρχουν στην παραγωγή και σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τα γεώμηλα σαν παράδειγμα. Είδαμε συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών στην εσοδεία των γεωμήλων. Ο Ολλανδός από το Βαχενίχεν. Ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις ε, απευθύνθηκαν ε, και σε μένα ή τουλάχιστον να προσπαθήσω να τις απαντήσω. Αφορούν το μέλλον της γεωργίας οι ερωτήσεις αυτές. Δύσκολα μπορεί κανείς να το προσδιορίσει, αλλά υπάρχουν μελέτες που μας δείχνουν διαφορά μεταξύ γεωργίας που στηρίζεται στην παραγωγή αφενός και της γεωργίας ε, που προσεγγίζεται ε, μέσα από την κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών. Είναι σημαντική προφανώς η γεωργία για την οικονομία. Αλλά υπάρχουν και άλλες ε, χρήσεις της. Πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα. Αυτό είναι σίγουρο και απαραίτητο. Ε, όταν υπάρχει προσαρμοστικότητα υπάρχει και μετριασμός. Οι προσπάθειες μετριασμού επικεντρώνονται στις ε, μεθόδους εντατικής γεωργίας ε, που διαφέρουν από την πολυλειτουργική γεωργία. Οι προσεγγίσεις διαφέρουν. Όσο πιο εντατική η γεωργία, ε, τόσο μεγαλύτερες ε, δυνατότητες υπάρχουν για παρεμβάσεις. Οι γεωργοί πρέπει να συμμετέχουν στην ε, προσαρμογή. Μπορεί να θέλουν με το άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς να έχουν και εκείνοι ένα μερίδιο παραγωγής ενέργειας. και στην κτηνοτροφία υπάρχει προσπάθεια να συμμετέχουν στις λύσεις Το θέμα της τεχνολογίας είναι σημαντικό. Υπάρχουν, αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται όμως με τον καλύτερο τρόπο. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, η παραγωγή σε θερμοκήπια είναι πολύ σημαντική, αλλά πάλι χρειάζονται επενδύσεις. Το θέμα δεν είναι εντατική ή εκτατική. Και τα δύο πρέπει να τα δούμε από την άποψη της αποτελεσματικής αποδοτικής οργάνωσής τους και βεβαίως αποτελεσματική χρήση ε, των πόρων, ασφάλεια τροφίμων. Εδώ έχουμε το 1α σενάριο ανοιχτή αγορά που εξαρτάται από τις παγκόσμιες τιμές, τις τιμές στις διεθνείς, στη διεθνή αγορά και πάλι οι επιπτώσεις στους μεμονωμένους γεωργούς εξαρτώνται από τα διαφορετικά σενάρια γιατί υπάρχει διαφορετικό σκεπτικό στο 1α και στο 2β. Οπωσδήποτε όλα αυτά πρέπει να δούμε σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Δεν θα μιλήσω για τις κλιματικές αλλαγές γιατί δεν είμαι ειδικό εκεί. Για το μετριασμό. Εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Η πολιτική της ε, γεωργικής διατήρησης είναι ο καλύτερος τρόπος και αυτό περιλαμβάνει και τα δάση, τους ε, φράχτες ε, και πολλά άλλα. Επίσης, όταν μιλάμε για άρρωση των εδαφών, η μηδενική άρρωση αποτελεί πολύ ενδιαφέρουσα μεθοδολογία. Όμως, δύσκολα μπορεί να ε, προσδιοριστούν ποσοτικοί δείκτες εδώ και υπάρχουν ε, και ε, παράμετροι που δεν είναι μόνιμες εδώ, που παίζουν ρόλο όταν μιλάμε για τη μέθοδο του οργώματος. και βέβαια πρέπει να δούμε τις γεωργικές πρακτικές ε, γιατί ορισμένες από αυτές ε, είναι, αποθαρρύνουν προς αυτές τις μορφές άρρωσης. Ευχαριστώ. Οι εμπειρογνώμονες από τον πρώτο γύρο θέλουν να παρέμβουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των υδάτων, σε ένα σύστημα καλλιέργειας όπου ο κύκλος του αζότου και του άνθρακα και του ύδατος συνδέονται μεταξύ τους. Και όταν ε, κάνουμε το όργωμα διαταράσσουμε και τους τρεις αυτούς κύκλους το νερό θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως από τα θέματα του άνθρακα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δέσμευση του άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης συνδέεται άμεσα με το νερό που καταναλώνεται. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο τέθηκε σε σχέση με το άζωτο και τα λιπάσματα. για να κάνουμε συνθετικά, τα συνθετικά λιπάσματα εκλείουν ένα τόνο διοξιδίου του άνθρακα στην, ατμόσφαιρα. Θα και πρωτοξίδιο του αζότου. Θα πρέπει να μάθουμε να δεσμεύουμε αυτό το άζωτο. Χρειαζόμαστε περισσότερα ψυχανθή κατ' ουσία. Έχουμε τον Τόμ Χίγκερ στι Ηνωμένε Πολιτείε που είπε ότι η βιολογική καλλιέργεια σφαιρικά θα υποστηρίξει ένα πληθυσμό 4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα έχουμε πάνω από 6,7 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Και ε, θεωρώ τα ζούχα λιπάσματα είναι σημαντικά για την ε, παραγωγή τροφίμων, αλλά ρηπαίνουν πάρα πολύ το νερό και έχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Έχουμε 70% ε, του εδάφους είναι νερό. Ε, στις υπάρχουν χορτολιβαδικές εκτάσεις και θα πρέπει να υποστηρίξουν τα εδάφη την αύξηση του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε πιο εντατικές καλλιέργειες στις αρωτρές γιες και θα πρέπει να αξιοποιούμε πιο αποτελεσματικά τους φυσικούς ε, πόρους για να το πετύχουμε. Ε, ε, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια αύξηση τροφίμων για αυτή την τον ταχαίως αυξανόμενο πληθυσμό. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές ε, που θα είναι πιο βιώσιμες. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ε, είναι η ομαδική εργασία. Νομίζω ότι χρειάζονται οι χρειάζονται οι πολιτικοί να συμβάλλουν οι καλλιεργητές και οι καταναλωτές. Όλοι αυτοί θα πρέπει να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα επισητιστικής ε, διατροφικής ασφάλειας. για να απευθυνθώ στην ερώτηση της κυρίας όσον αφορά την ε, αντίσταση στην αποδοχή της μη άρρωσης. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση για τους καλλιεργητές. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι εδώ, αρχικά, κάποια ρίσκα, αλλά αυτή τη στιγμή οι καλλιεργητές ευθύσουν αυτό το νέο σύστημα, θα σταθούν πιο άνετα μέσα σε αυτό. Αφορά, ε, όλα αυτά είναι πολιτιστικά θέματα, ζητήματα ε, πρόσληψη των νέων μοντέλων και ερμηνεία. Το βασικό εμπόδιο βεβαίω είναι η άρνηση να αλλάξουν κάποιε νοοτροπίε. Ε, υπάρχουν ανησυχίες για άσκηση κριτικής από τους άλλους κλπ. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες που προϋποθέτουν νέο εξοπλισμό και ένα υψηλό επίπεδο διαχείρισης. Ε, νομίζω ότι δεν είναι κακό να βελτιώσουμε τις διαχειριστικές μας ικανότητες. Ένα άλλο στοιχείο είναι οι επιδοτήσεις της ε, Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Η, η δική μας ε, χρειάζεται να επιδοτήσουμε την, τις βιολογικές καλλιέργειες και τα οικοσυστήματα τα οποία θα είναι πιο βιώσιμα και νομίζω ότι έχει κρίσιμη σημασία να το πράξουμε. Κανείς δεν θέλει να μιλάει για τον έλεγχο του πληθυσμού αλλά οι πόροι μας είναι πεπερασμένοι και αν δεν τους αξιοποιήσουμε παρκώς αυτό θα είναι εις βάρος του πληθυσμού και του πολιτισμού μας. Ευχαριστούμε πολύ τους εμπειρογνώμονες και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Στεφάν Λεφόλ για, τις, ε, για τα τελικά του συμπεράσματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ όπως και εσείς θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που ακούσαμε σήμερα το πρωί γιατί ήταν ξεκάθαροι σχετικά με τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και πρότειναν αρκετές λύσεις. Alors je voudrais juste lever un euh, για τους σκεπτικιστές σχετικά με τις κλιματολογικές αλλαγές. Πάντα ε, υπάρχει σκεπτικισμός όταν τίθεται ένα ερώτημα. Αλλά όπως ε, ακούστηκε υπάρχουν πια κάποια αντικειμενικά στοιχεία. Αν πάτε στον ειρηνικό, ο κόσμος που ζει σε μικρά νησιά βλέπει η θάλασσα να τους απειλεί. Αν πάτε στον Μπαγκλαντές ε, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις γιατί και εκεί από ό,τι φαίνεται υφίστανται τις συνέπειες των, της πλημμύρες. Αν δείτε τι συμβαίνει στην Ισπανία σαν παράδειγμα και το είπε ένας εμπειρογνώμων, οι θερμοκρασίε αυξήθηκαν και η ξύρανση γενικά των γεών είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ότι δεν τρέχει τίποτα και η αναφορά στους δεινοσαύρους που έγινε από τον αντιπρόεδρο είναι ότι οι δεινόσαυροι δεν κατάλαβαν τι τους περίμενε, ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Και εμείς ακριβώς επειδή είμαστε οι διάδοχοί τους πρέπει να δούμε αν θα κάνουμε σαν τους δεινοσαύρους. Θα κάνουμε δηλαδή ότι δεν συμβαίνει τίποτα και κάποια στιγμή θα εξαφανιστούμε ή θα προσπαθήσουμε να προστατευτούμε γιατί η γη θα συνεχίσει να γυρνάει είτε είμαστε εμείς επάνω είτε όχι. Λοιπόν, έτσι τίθεται το πρόβλημα. Η κυρία Μαγκίνε είπε ότι πέρα του θέματο αυτού, και οι σκεπτικιστές θα επιμείνουν έτσι και αλλιώ, τέθηκε το θέμα της υπερθεύμανσης του πλανήτη και της αντιμετώπισης των συνοπιών της υπερθεύμανσης αυτής, συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο θα παράγουμε στη γεωργία σε υψηλό επίπεδο με μεγάλη ποικιλία, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση και διατηρώντας τους σπόρους που βρίσκονται στη βάση της παραγωγής. Η γεωργία είναι ο κατεξοχήν κανόν, τομέας, ο οποίος είναι σε επαφή, θα έλεγα, με ό,τι ζωντανό υπάρχει πάνω στη γη, και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την προσπάθεια διαμόρφωσης νέων σχημάτων στο μέλλον που θα διασφολήσουν την αηφορία της προσπάθειάς μας να δώσουμε απαντήσεις μάλιστα στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Είχα θέσει ένα ζητούμενο. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε πρέπει να είναι σφαιρική. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά με οδηγίες αυτόνομες η μία από την άλλη. Ένας από τους εμπειρογνώμονες είπε ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ελκυστικά ε, ικανοποιητικές μάλλον για τους γεωργούς αλλά και για την κοινωνία και για το λεγόμενο κοινό αγαθό, δηλαδή για τη διασφάλιση του πλούτου των φυσικών πόρων, της βιοποικιλομορφίας και επαναλαμβάνω το θέμα των νερών, του ύδατος, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, ακούσαμε για τη διατήρηση του εδάφους, για την διαχείριση των δασών, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην συγκράτηση του άνθρακα στο έδαφος και εγώ θέλω να υπάρξει θέμα και για τα δάση, η βιομάζα από τα δάση είναι αναπόσπαστο κομμάτι και πρέπει να είναι της ευρωπαϊκής πολιτικής και ταυτόχρονα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ε, για τον τρόπο με τον οποίο η κοινή αγροτική πολιτική μπορεί να μας επιτρέψει να πετύχουμε αυτήν την μετάβαση την οικολογική αν θέλετε. Ένα πράγμα είναι να κάνουμε τη διάγνωση, ένα πράγμα είναι να κάνουμε τη διαπίστωση συνέπεια των ε, επιλογών που έχουμε κάνει στα πλαίσια της παραδοσιακής συμβατικής γεωργίας και ένα άλλο πράγμα να δούμε πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες μας στο μέλλον γιατί οι πολίτες θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα της γεωργίας και της κοινή γεωργικής πολιτικής μόνο αν μπορέσουν να τους δώσουμε σφαιρικότερες απαντήσεις γύρω από το μέλλον του πλανήτη. Γι' αυτό ακριβώς η συζήτηση είναι βασική. Τώρα ξεκινάει βέβαια, εμείς ανοίγουμε προοπτικές και τις συνδέουμε τις προοπτικές αυτές με τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2013. Χαίρομαι για τη συζήτηση που προηγήθηκε σήμερα το πρωί και το μόνο το οποίο εύχομαι είναι να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε νέες επιλογές στη Γεωργία και ιδιαίτερα νέες επιλογές από τη Γεωργία στην κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Οδηγούμεθα πλέον στο τέλος της ακροάσεώς μας. Έχω και εγώ την εντύπωση ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η ακρόαση αυτή, ιδιαίτερα καρποφόρα. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα θα μας επιτρέψουν να εκμεταλλευτούμε σωστά την έκθεση την οποία συνέταξε ο συνάδελφος Λεφόλ. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου, 12η μεσημβρινή και η ψηφοφορία.